Dear colleagues, I would like to start the meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν έχουμε λάβει κάποιο αίτημα τροποποίηση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Επομένω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Να σα ενημερώσω τη συνεδρίαση ω συνήθω αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Να περάσουμε στο σημείο 3 τη σημερινή της διάταξη, ε, έγκριση των πρακτικών, της συνεδρίασης, τη 23η, 24η Ιανουαρίου και 19 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά έχουν διατεθεί, έχουν διανεμήθει. Αν δεν έχετε αντίρρηση, αν δεν εκφραστεί κάποια αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνουν τα πρακτικά στο τέλος της σημερινής συνεδρίασής μας. Έχω κάποιες ε, ανακοινώσεις ε, μετά την τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν είχαμε χρόνο να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές. Καταρχήν, μια ενημέρωση για το τι πράξαμε στη γραπτή διαδικασία, κατανομή γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων σε συγκεκριμένους συναδέλφους, ε, κ. Σταυρακάκης, προϋπολογισμός 2014, κατόπιν κ. Φραγκούτ, για το άνοιγμα των αγορών, για τις ε, ε, υπηρεσίες μεταφοράς επιβετών στους σιδηροδρόμους, επίσης για τις μεταφορές για τον ενιαίο χώρο σιδηροδρόμων, Μαρία Τερέσα Σάνσα Σμίτ για το σιδηροδρομικό σύστημα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις, έχουμε Καρίν Κάντερμπαχ με έκθεση δίας πρωτοβουλίας για το πόσο η Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στο να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις startups για τη δημιουργία θέσεων εργασία και έκθεση πρωτοβουλίας ε, για την ανεργία των νέων. Θα πάει στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, δεν ξέρουμε ακόμη σε ποιον, δεν έχουμε το όνομα και καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της θητείας έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την κατανομή εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας για ε, το θέμα των σλότ των χρονοθερίδων. Και θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η απόφαση στην προηγούμενη συνεδρίαση των συντονιστών του Φεβρουάριο ελήφθη. Αποφασίσαμε ότι από σήμερα μέχρι τα τέλη της ε, θητείας μας ε, θα έχει κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες αναλάβει μία έκθεση της πρωτοβουλίας ανάλογα με το πώς θα λειτουργούν οι ποσοστώσεις και επίσης συμφωνήσαμε ότι θα ζητηθεί άδεια για τις τέσσερις εκθέσεις βάσει των προτάσεων που θα έρθουν από το ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές, τους Πρασίνους και το ΕΣΥΑΡ. Και κατόπιν, ε, σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία, συμφωνήθηκε από τους συντονιστές ότι η πρώτη ομάδα, το πρώτο μπλοκ εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας αποτελείται από μια έκθεση από το ΕΛΚ για την ευφύ εξειδίκευση από τους σοσιαλιστές για την ετοιμότητα των κρατών μελών για την ε, κατάλληλη έναρξη της πολιτικής συνοχής, το ECR για την περιφερειακή πολιτική συνοχή, ίσως ε, ε, σχέδιο κρατικής υποστήριξης, επίσης να ζητήσουμε έγκριση για μια τέταρτη έκθεση από τους Πρασίνους για τα φιδίκτια. Θα συζητηθεί επίσημα τον Απρίλιο, όταν θα ψηφίσουμε την έκθεση του κ. Γκάιτς. Που πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Και επίσης το Φεβρουάριο συμφωνήσαμε ότι η φιλελεύθερη Κικούε θα παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις για τις δικές τους αντίστοιχες εκθέσεις ιδίες, πρωτοβουλίες και κατόπιν λάβαμε αντίρρηση από τους ελευθέρους ότι δεν υποστήριξαν αυτή τη συμφωνία και θέλουμε να δουν την πρόταση στο πρώτο μπλοκ. Αυτά σε σχέση με τις συνεδρίες του Φεβρουαρίου. Θα σας αναφέρω και τα υπόλοιπα μετά τη σημερινή συνεδρία των συντονιστών. Αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ως έκθεση της συνεδρίας των συντονιστών. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο σημείο 4 της ημέρας της που σχετίζεται με την έκθεση Γιάννης Γκάιερ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Αλλά σήμερα έχουμε και την παρουσίαση της ε, μελέτης ε, για ε, τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ακούσουμε τον κύριο Τέντλσεν Χόφερ την κυρία Τέντλισεν Χόφερ που είναι διευθύντρια της ΜΕΤΙΣ στη Βιέννη και θα παρουσιάσουμε λοιπόν αυτή την έκθεση και θα τη συζητήσουμε. Η παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Τέντλινγκ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καλή... Καταρχήν να στήσω συγγνώμη. Πάντα ε, μου φαίνεται περίεργο να κάνω μια παρουσίαση σε ένα κοινό ε, το οποίο βλέπει την πλάτη μου, αλλά τι να κάνω. Ε, θα μείνω εδώ. Καλά, ένα λεπτό. Ο Μικέλ μου ζητάει να τονίσω ότι ε, ε, ε, δίνουμε ιδιαίτερη μεταχείριση στην κυρία Τότλινγκ, απλά ήθελα να το πω. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω ένα έγγραφο το οποίο έχει να κάνει με τις περιφερειακές στρατηγικές για βιομηχανικές περιοχές και μάλιστα παλαιές βιομηχανικές περιοχές και πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να επανερχόμαστε στις περιοχές. Εγώ όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο ε, με το θέμα των παλαιών βιομηχανικών περιοχών. Ήταν το σημαντικότερο θέμα ε, στην περιφερειακή πολιτική τότε, αλλά κατόπιν έφυγε από τη μόδα. Η ενημέρωση, το έγγραφο λοιπόν αυτό, το οποίο είμαι το έχετε διαβάσει όλοι σας, με τι ασχολείται. Καταρχήν, με τις προκλήσεις της διαρθρωτικής μεταμόρφωσης των περιοχών αυτών και έχοντας ιδιαίτερα κατά νου τις παλαιές βιομηχανικές περιοχές. Το δεύτερο ερώτημα είναι η πολιτική συνοχή σε πώς μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία αυτή και θα σας το περιγράψω αυτό με τέσσερα νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα παραδείγματα με τις πόλεις Μάνσεσταρ, Έσεν, Λίλ και Μπιλμπάο είναι και οι τέσσερις πόλεις που είχαν τεράστιες ανάγκες ε, ε, για διαρθρωτική αλλαγή και είναι ακόμα ζωντανές παρότι έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Η αναδιάρθρωση στις πόλεις αυτές ε, φυσικά πραγματοποιήθηκε και με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων και θα ε, καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα για τις πολιτικές συνοχής ε, και κάποιες επικρίσεις ενδεχομένως για την πολιτική συνοχή, που είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλειστικά αφιερωμένη στην έξυπνη εξειδίκευση και φαίνεται να ξεχνά τις άλλες πτυχές. Το πρώτο θέμα λοιπόν, ε, πρωτού μιλήσω για τις παλαιές βιομηχανικές περιοχές. Ε, εδώ βλέπετε μια σύνοψη την οποία μόλις ε, σας περιέγραψα. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια να αναφερθώ στις να στη σημασία της βιομηχανίας, διότι η βιομηχανία Παρότι ε, έχει συζητηθεί πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωση λόγω της ε, οικονομικής κρίσης ε, και παρά την πρόσφατη παρακμή συνεχίζει να είναι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξη και αλλαγή. αλλαγής. Ήταν και στο παρελθόν και συνεχίζει να είναι. Αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ και συνεχίζει να διατηρεί πολύ σημαντικό επίπεδο όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Από ε, τις 100 ε, θέσεις που δημιουργούνται στη βιομηχανία δημιουργούνται 60 με 200 ε, στο υπόλοιπο της οικονομίας και αντιπροσωπεύει η βιομηχανία το 80% των εξαγωγών καθώς και το 80% των ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και ανάπτυξη. Η βιομηχανία λοιπόν ήταν ο κινητήρας της ε, κοινωνικής, πολιτιστικής ε, και οικονομικής ανάπτυξης, ε, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Έχει αυξήσει δραματικά την παραγωγικότητα, την καινοτομία. Έχουμε διάσπαση της αλυσίδας παροχής και η εικόνα των ε, καπνοδόχων που βγάζουν ε, καπνό ε, ανήκει στο παρελθόν πια. Έχουμε τώρα αναπροσανατολισμό του εργατικού δυναμικού και έχουμε πολύπλοκες αλυσίδες αξιών τώρα πια. Έχει αλλάξει λοιπόν σημαντικό τρόπο που παράγονται τα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της κρίσης έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κάτι που αντιπροσωπεύει το 10% του ε, εργατικού δυναμικού. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανάκαμψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την βασίσουμε στην πραγματική οικονομία, στην παραγωγή δηλαδή και η εμβληματική πρωτοβουλία για την βιομηχανική πολιτική, την ενίσχυση του ανταγωνισμού ε, ε, απαιτεί ε, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανία και ιδιαίτερα αναφέρεται στην πολιτική συνοχή και στο πρόγραμμα πλαίσιο. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για πιο ε, ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία για οικονομική ανάκαμψη ε, απαιτεί μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση, κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι απαιτεί ε, μετακίνηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω νέων κατασκευών, κάτι που θα οδηγήσει και σε νέες απαιτήσεις, αύξηση της συζήτησης. Ε, αλλά είναι απόλυτα ασαφές τι ακριβώς είναι η, βιομηχανία. Φαντάζομαι ότι όλοι από εσά έχετε ε, μια εικόνα ε, εργοστασιακών καπνοδόχων, αλλά η βιομηχανική πολιτική είναι κάτι που απευθύνεται στη βιομηχανία και αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι η Eurostat θεωρεί ότι είναι ο, ο ε, τομέας ε, ε, παραγωγής προϊόντων. Κάποιοι συμπεριλαμβάνουν εδώ και κάποιες υπηρεσίες. Η βιομηχανία λοιπόν είναι μια καποστολή εικόνα. Βιομηχανικός τομέας είναι ο τομέας που παράγει. Ελπίζω να μην σα προκαλεί σύγχυση ο πίνακα που βλέπετε. Θέλω να ξεκινήσω στα δεξιά, κάτω δεξιά. Τι είναι η βιομηχανική πολιτική. Ε, είναι κάτι που βρίσκεται στις ρίζες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε τη δεκαετία του 50. Το πρόβλημα ήταν να ξεπεραστούν ε, τα προβλήματα στον ε, τομέα χάλιβα και άνθρακα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν συνεργάστηκαν για να ε, λύσουν το πρόβλημα των ε, βιομηχανιών τους που βρισκόντουσαν σε παρακμή. Ε, σε εθνικό επίπεδο ενθάρρυναν τις, τους νέους παραγωγικούς τομείς αλλά συνεργάστηκαν για να καταπολεμήσουν τα προβλήματα στις, στους τομείς που τότε έδιαν. Ε, έχουμε λοιπόν την οριζόντια προσέγγιση που περιλαμβάνει την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες, ε, τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς κλπ. Και επίσης έχουμε το γενικότερο πλαίσιο, την καλύτερη ρύθμιση, την κρατική ιδιοκτησία κλπ. Ε, περιλαμβάνονται λοιπόν εδώ οι συνθήκες πλαίσιο και οι οριζόντιες πολιτικές καθώς και οι τομεακές πολιτικές οι οποίες Τώρα πια είναι ομαδικέ ενοποιημένε τομεακέ πολιτικέ. Αυτέ οι πολιτικέ δεν είναι οι μόνε που επηρεάζουν την ε, βιομηχανία. Ίσως η χρήση τη γη ή ε, η η νομοθεσία να επηρεάζει περισσότερο την ε, βιομηχανία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλέ πολιτικέ που δεν απευθύνονται άμεσα στον τομέα της βιομηχανίας, που όμω μπορεί να την επηρεάζουν περισσότερο. Η βιομηχανική πολιτική εξορισμού είναι μη εδαφική πολιτική. Ωστόσο, πραγματοποιείται σε μεγάλο, ε, ε, ε, εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κάποια εδάφη και βλέπετε στις παλιές βιομηχανικές περιοχές πώς εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Ε, έχουμε λοιπόν ε, την παλιά βιομηχανία άνθρακα και χάλιβα, την, ε, την κλωστοϊφαντουργία κλπ. Οι παλιές ε, βιομηχανίες λοιπόν όταν βρέθηκαν υποπίεση λόγω της ανακατονομής εργασίας σε διεθνές επίπεδο η παραγωγή αυτή μεταφέρθηκε σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι περιοχές λοιπόν αυτές αντιμετώπισαν πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία Ε, ήταν ε, αρκετά σοβαρά τη δεκαετία του 1970. Έγιναν τότε αρκετές μελέτες οι οποίες ανέλησαν ε, την, τις διάφορες εξαρτήσεις και τις οδούς προς την αποκατάσταση των περιοχών. Είναι σαφές για ποιες περιοχές μιλάμε. Μιλάμε για την βορειοανατολική Αγγλία, την περιοχή Ρουρ, την χώρα των Βάσκων Ε, καθώς και κάποια μέρη των νέων κρατών μελών, ε, στα οποία όμως δεν έχει δοθεί μεγάλη ε, προσοχή. Αντιμετώπιζαν λοιπόν οι περιοχές αυτές ίδιου τύπου προβλήματα, αλλά ίσως κάπως αργότερα, προβλήματα τα οποία παραμελήθηκαν από τα καθεστώτα τους πριν πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Οι νέες προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ένωση μας κάνει να παραμελούμε τα παλιά προβλήματα, Όπω είναι η διεύρυνση ε, προ τα ανατολικά, ε, η λισαβονοποίηση τη πολιτική συνοχή, η οικονομική κρίση, καθώ ε, και η έλλειψη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Για να μην έχετε απλά μια θεωρητική εικόνα των όσων συμβαίνουν, έχουμε εξετάσει τέσσερις περιπτώσεις. Μιλάμε κυρίω για αστικέ περιοχές που αντιμετωπίζουν ε, τα προβλήματα αυτά, διότι οι βιομηχανικές περιοχές εξορισμού είναι αστικές. Πώς λοιπόν ε, τα κατάφεραν ε, οι διάφορες περιοχές στη διαδικασία της μετατροπής. Έχουμε λοιπόν την πόλη Έσεν της Γερμανίας, την Έση, στην περιοχή Ρουρ, την Λίλ, στη Γαλλία κοντά στα βελγικά σύνορα, το Μάντσεστερ που είναι το, το της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη ε, και το Bilbao. που μεγάλωσε κυρίως λόγω των ορυχείων, ε, αλλά κατόπιν επεκτάθηκε και ε, στα ναυπηγεία. Πίσω από τις πόλεις αυτές υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της Ευρώπης, ε, αλλά 20 ε, λεπτά πρέπει να μιλήσω, οπότε μάλλον δεν ε, θα έχω το χρόνο να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες για τις πόλεις αυτές. Νομίζω πάντως ότι δίνουν πολύ, καλό, πολύ καλή εικόνα του πώς εξελίχθηκε η Ευρώπη και τι ακριβώς είναι η εδαφική ανάπτυξη. Αυτές οι τέσσερις πόλεις Ε, είναι παραδείγματα πόλεων ε, που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα. Ε, τι κοινό έχουν. Έχουν περιοχές μολυσμένες με παλιά υποδομή. με παλιά εργοστάσια και παλιά κτίρια. Έχουν κατοικίες οι οποίες χρήστηκαν για πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό φτωχής, κακής ποιότητας έχουν μη ελκυστικούς δημόσιους χώρους, ποτάμια και ανοιχτές περιοχές που ε, να αναδιαρθρωθούν. Θυμάμαι πρώτη φορά που επισκέφθηκα την περιοχή Ρουρ, ε, υπήρχαν ακόμα ανοιχτοί υπόνομοι, κάτι απίστευτο για τη δεκαετία του 70. Τέτοιου τύπου προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουν οι περισσότερες από αυτές τις πόλεις. Οι τέσσερις αυτές πόλεις με εντυπωσιακό τρόπο κατάφεραν να αλλάξουν από παλιές παραμελημένες περιοχές σε λίγο πολύ ε, ε, ανεπτυγμένες πόλεις. Και να σας δείξω λίγο τα παρασκήνια, πώς κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Και το βασικό μου μήνυμα είναι ότι χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά δεν χρειάζονται μόνο χρήματα. Καταρχήν, αυτά που σας περιέγραψα πριν, ε, την ε, ε, ανακαίνιση των κατοικιών, την ανοικοδόμηση της υποδομής, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μια τοπική αρχή ή εθνική αρχή, όλα αυτά απαιτούν συνεργασία και οι τέσσερις αυτές περιοχές έχουν επιδείξει πολύ σημαντικά παραδείγματα συνεργασίας στην περιοχή Ρουρ. Νομίζω ότι έχουμε την παλαιότερη ένωση χωροταξικής, ε, χωροταξικού ε, προγραμματισμού και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο διακυβέρνησης, διότι πριν 30 χρόνια νομίζω ή μπορεί και περισσότερο, μια σειρά τοπικών αρχών ανέθεσε την αρμοδιότητα ε, για χωροταξικό προγραμματισμό σε μια ένωση που τώρα έχει αποκτήσει και συνέλευση όπου συμμετέχουν οι ε, τοπικές αρχές και περιφέρειες και περιφερειακές αρχές. Στη ΛΙΛ το θέμα της ε, διασυνοριακής συνεργασίας επίσης ήταν πολύ σημαντικό και η περιοχή ανάμεσα στη Γαλλία και στο Βέλγιο δεν είναι ακριβώς ένα φυσικό σύνορο, ε, είναι λίγο πολύ το ίδιο τοπίο. το σύνορο απλά μια γραμμή είναι, ένα εμπόδιο. Και η μακρά διαδικασία συνεργασίας ε, ολοκληρώθηκε με μια EGTC ε, με την ε, περιοχή Lille Κόρτρεϊκ Τουρνέ που αποτελεί καινοτομία στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα μπορούσα και για τις άλλες δύο πόλεις να σας δώσω παραδείγματα οριζόντιας συνεργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητάμε τη διακυβέρνηση, διότι η διακυβέρνηση δεν είναι μόνο ε, διακυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, έχει να κάνει και με την ε, οριζόντια συνεργασία. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα στο Πιλπάο. Ε, δημιουργήθηκαν ενώσεις που συνδύασαν ε, ε, χρήματα από το τοπικό, ε, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με ιδιωτικού πόρου. Και τρίτον, χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στον προγραμματισμό, την οικονομική ανάπτυξη, την αγορά εργασία και οι τέσσερις αυτές πόλεις έχουν αποτελέσει πολύ σημαντικά παραδείγματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι η εργάσια συνεργασία, το άλλο είναι ο συνδυασμός ε, τοπικού και εθνικού επίπεδου, ε, τοπικής και εθνικής προσέγγισης. Τελικά δεν υπάρχει κάποια συνταγή, αλλά Ε, μιλάμε για ε, κάποια περιοχή που να μπορεί να επωφεληθεί από την τοπική και εθνική προσέγγιση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν είχε προγράμματα ανάπτυξης για τι περιοχές, αλλά προσπάθησε να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες. Το Μάντσεστερ απέκτησε κάποιες ε, νέες βιομηχανίες ε, μέσα από μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης εθνικού επίπεδου. Είχαμε λοιπόν μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και προσέγγιση μέσω της τεχνολογίας. Στην ΕΣΥ Ε, ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα που είχαμε ήταν ε, η ε, είχαμε την σημαντική έκθεση κτηρίων το πάρκο Ιμπα Έμσερ που ξεκίνησε καταρχήν από την ανακαίνιση παλιών βιομηχανικών κτηρίων και την μετατροπή τους σε κάτι καινούριο και δημιούργησε πολλά επιμέρους προγράμματα ε, πάνω σε κτίρια. Η Λίλη είχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, είχε εθνική πολιτική για ε, αποκέντρωση ε, και οι αποκεντρωμένες περιοχές αποτέλεσαν πόλους τεχνολογίες. Και στο Μπιλμπάο είχαμε συμπράξεις δημοτικού και, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Πέντε λεπτά μου δίνεται ακόμα. Ε, ωραία, τότε δεν θα μιλήσω για τις επιτυχημένες στρατηγικές. Ε, τι μπορεί να κάνει η πολιτική συνοχή. Ε, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει ε, τα πάντα. Πολύ λίγοι είναι οι περιορισμοί, αλλά... Δεν θα αναφερθώ σε αυτά, διότι μπορείτε να τα διαβάσετε στην, στο, έγγραφο, το πώς οι διάφορες πολιτικές συνέβαλαν στην ανάπτυξη στο Bilbao, το Manchester και ε, την ΕΣΥ. Ήταν ουσιαστικά εμβληματικά προγράμματα ε, ε, και βιομηχανική αναδιάρθρωση. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Καταρχήν, και θέλω να το τονίσω αυτό στα τελευταία πέντε λεπτά που έχω, η βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να ξαναμετατρέψει βιομηχανικές ε, περιοχές. Ένα από τα μαθήματα που ε, ε, έχουμε από τη βιομηχανική πολιτική της δεκαετίας του 50, 60 και 70 είναι ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις υπερτιμούν τον κίνδυνο της τις αποτυχίες ε, στην αγορά και υποτιμούν ε, την ε, δυνατότητα αποτυχίας των δικών τους κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ουσιαστικά δηλαδή προτιμούν πεπαλαιωμένες προσεγγίσεις. Αλλά μια διαφοροποιημένη οικονομία συνδυάζει διάφορες βιομηχανίες και έτσι τελικά πετυχαίνει. Οι βιομηχανικές στρατηγικές ε, λοιπόν είναι επικίνδυνες ε, εάν ε, ευνοούν τους ισχυρούς στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, αν κανείς θέλει να ευνοήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. Η βιομηχανική πολιτική λοιπόν θα πρέπει να ε, στηρίξει την ε, διεθνή ανταγωνιστικότητα, ενώ η ε, πολιτική συνοχή θα πρέπει να βοηθήσει τις πόλεις και τις περιοχές να βρουν τον σωστό τρόπο προς την αποκατάσταση και ανάκαμψη. Σημαντικότερο είναι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι στρατηγικές να προωθήσουν διαφοροποιημένη ανάπτυξη, δηλαδή να μην επικεντρωθούν αποκλειστικά στην έρευνα και τεχνολογία, διότι Και δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Αλλά εάν η πολιτική συνοχή ε, ε, ε, προσανατολιστεί προς την έρευνα και τεχνολογία, είμαι πεπισμένη ότι οι βιομηχανικές περιοχές θα, θα βρεθούν σε πιο αδύναμη θέση. Διότι Οι επενδύσεις σε περιοχές που αναπτύσσονται αποφέρουν περισσότερα από ότι οι επενδύσεις σε περιοχές που έχουν σημαντικές ανάγκες. Και καθότι δεν υπάρχει εδαφική προσέγγιση, καταρχήν ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, εξετάσουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα και πώς επωφελούνται οι διάφορες περιφέρειες, διότι εμείς ε, πήραμε τα, το υλικό από διάφορες πηγές χωρίς ε, να γνωρίζουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα και πιστεύουμε ότι οι παλιές βιομηχανικές περιοχές που βρίσκονται στον δρόμο προς την ανάκαμψη και τον ε, ε, αναπροσανατολισμό συνεχίζουν να χρειάζονται χρήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, το χρήμα δεν είναι τα πάντα. Ε, αυτό που λείπει από την πολιτική συνοχή είναι μια πραγματική και ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση. Δεν ε, απαγορεύεται αυτό στους κανονισμούς, αλλά ούτε απαιτείται. Και να σας δώσω παράδειγμα του Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης, που έχει μια μακρά παράδοση τοπικής ανάπτυξης. Το Λίντερ. ναι. Ναι, το Leader. Έχει λοιπόν καθιερώσει μια εδαφική προσέγγιση, ε, αλλά πιστεύω ότι με ολοκληρωμένες ε, ε, εδαφικές επενδύσεις στο νέο κανονισμό Υπάρχει δυνατότητα να οριοθετήσει κανείς μία περιοχή και να εφαρμόσει διάφορα πακέτα δράσεων. Ωστόσο, από όσα έχω ακούσει, φαίνεται ότι το ότι ο περιορισμός σχετικά με το 5% ε, δεν θα επιβιώσει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που πραγματικά απαιτείται για την πολιτική συνοχή είναι οι παλιές, βιομηχανικο... οι βιομηχανικές περιοχές να στηρίξουν και να προσελκύσουν ε, οριζόντιες και εγκάρσεις συνεργασίες ώστε να υπάρχουν σχέδια ε, τοπικής ανάπτυξης για τις περιοχές αυτές, ώστε να μπορέσουν να αποφεληθούν και αυτές από το πρόγραμμα. Σε πολλά κράτη-μέλη, σε επίπεδο πιο χαμηλό από ε, το περιφερικό πρόγραμμα, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης ε, σχεδίου δράσης ή κοινής στρατηγικής. Πιστεύω λοιπόν ε, ότι αυτή η μέθοδος ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ε, θα μπορέσει να ε, ξαναβρει μια θέση στο χάρτη για τις παλιές βιομηχανικές περιοχές και να επιστήσει την προσοχή του κόσμου στα προβλήματα και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την συνεργασία και όχι μόνο τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ. Θα γίνει μετά συζήτηση. Θα αρχίσουμε ίσως από την Κωνσταντσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ να ε, απαντήσω σε κάποια από τα πράγματα που μόλις παρουσιάστηκαν. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσω από τα speaking notes που μου έδωσε ο εισηγητής, από τις σημειώσεις που μου ε, ε, έδωσε ο εισηγητής. Σήμερα λοιπόν έχετε το σχέδιο μιας έκθεσης στα εγγραφά σας που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στο έγγραφο εργασίας. γίνονται διάφορε εκκλήσει προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη σχετικά με το πώ μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των παλιών βιομηχανικών περιοχών. Το σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει έναν κατάλογο των σημαντικότερων ε, προκλήσεων για τις ε, πρώην βιομηχανικές περιοχές ε, και ο κατάλογος αυτός που υπάρχει και στην ε, μελέτη. Νομίζω ότι, μάλλον συγγνώμη, ο κατάλογο αυτός νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στον κατάλογο που υπάρχει στη μελέτη αυτή. Το σχέδιο έκθεσης ε, τονίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα των ε, βιομηχανικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη περίοδο ανάπτυξης και σύντομο χρονικό διάστημα ε, συρρήκνωσης ε, της ε, βιομηχανικής ανάπτυξης και την ανάγκη αναπροσανατολισμού. Το σχέδιο έκθεσης δείχνει ότι οι θέσεις αυτές δεν, βρίσκονται σε μάλλον μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλες περιοχές όσον αφορά τις, την αναγνώριση των αναγκών αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο έκθεσης επίσης αναφέρει ότι και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπάρχουν δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη ε, που ε, ε, συχνά όμως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των περιοχών αυτών. Για την ανάπτυξη λοιπόν τέτοιων περιοχών θα πρέπει να αναπτύξουμε σχέδια που προτείνουμε ως προϋπόθεση για την μελλοντική ε, πολιτική συνοχή, ώστε να έχουμε όσο γίνεται αποτελεσματική χρήση των ε, πόρων. Το σχέδιο έκθεσης ε, καλεί τα κράτη-μέλη να αποφύγουν ιδιαίτερα πολύπλοκους κανόνες ε, για τους ε, παραλήπτες ε, των πόρων και είναι απόλυτα σαφές ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη έχουμε προσπαθήσει να απλοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να πραγματοποιηθεί και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ο εισηγητής ε, στην έκθεσή του καλεί την ε, Κομισιόν να ε, αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση των βιομηχανικών περιοχών και να δει ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις ώστε σε διαπραγμάτευση, σε συζητήσεις με τις περιοχές να αναπτυχθούν περιφερειακές στρατηγικές. Όπως είπατε και στο μέλλον το, η αρχή ε, του προγράμματος LEADER θα χρησιμοποιηθούν ε, όχι μόνο για την ε, γεωργική ανάπτυξη αλλά και για τις αστικές περιοχές. Ο εισηγητής λοιπόν πιστεύει ότι υπάρχει εδώ μια ιδιαίτερη ευκαιρία για τις βιομηχανικές περιοχές. Η ευφυής εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική έννοια για τις βιομηχανικές περιοχές και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην ε, έκθεση, αλλά τελικά ε, δεν βρήκε χώρο ο εισηγητής στην ε, έκθεσή του. Ο εισηγητής αυτά μου ζήτησε να πω, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποιες δικές μου παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι με τη νέα προσέγγιση της διαθροτικής πολιτικής για τα επόμενα πέντε χρόνια ακολουθούμε έναν δρόμο τον οποίο θα έπρεπε να έχουμε ακολουθήσει ήδη πριν 7 χρόνια. Ε, πολύ καιρό πιστεύαμε, υπερβολικά πολύ καιρό πιστεύαμε ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητη η βιομηχανία. Ε, αυτή όμως είναι μια πολύ λανθασμένη αξιολόγηση και σίγουρα έχουν καταστραφεί στο μεταξύ πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ε, επιδιορθωθούν ε, ε, από ότι αν ε, δεν ε, είχαν καταστραφεί. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκαταστήσει κανείς μια βιομηχανική περιοχή από το να χτίσει μια καινούρια. Ξέρετε ότι προέρχομαι από την Ανατολική Γερμανία, στην Σαξονία, Σαξονία Σαξονία-Άνχαλτε και Θουρίνγκη και, και Θουρινγκία. Έχουμε Ε, σημαντικές ε, περιοχές ε, πρώην βιομηχανικές που είχαν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό αλλά είχαμε πολύ σημαντικές προσπάθειες ανοικοδόμησης. Κάτι που ίσως δεν έγινε με εξίσου εντατικό τρόπο σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Οπότε έχουμε την προσέγγιση ότι ναι, η νέα διαφορετική πολιτική σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και η ε, και υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα με την διορθωτική πολιτική. Γι' αυτό στις ε, διαπραγματεύσεις ε, δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τον τομέα των μετατροπών και την σχέση των βιομηχανικών περιοχών με την έρευνα και την τεχνολογία. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον σύνδεσμο αυτών διότι έτσι μπορούμε να έχουμε αναβιομηχανοποίηση, αναδιάρθρωση και ελπίζω κατά την ανάγνωση της μελέτης να βρω και κάποιες προτάσεις σχετικά με το τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σημαντικό είναι όμως να Μην θεωρούμε ότι η βιομηχανία είναι κάτι εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, είναι φθηνότερο εργατικό δυναμικό και δεν χρειάζεται να τηρούμε τις περιβαλλοντικές ε, ε, τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το θέμα της βιομηχανίας και με τη νέα διαρθρωτική πολιτική νομίζω ότι προωθείται ακριβώς αυτό. Αυτές λοιπόν ήταν οι παρατηρήσεις μου καθώς και οι παρατηρήσεις που μου έδωσε ο Γιάννης Γκάιερ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Κωνσταντσα από τους Κιώδης τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσκεκλημένη μας για την παρουσίασή της. Μας θύμισε κάτι που, στο οποίο επιμένουμε και εμείς πολύ τη λέξη μέλλον. Και εμείς το μέλλον θέλουμε να προετοιμάσουμε. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε πια τις παλιές μεθόδους του παρελθόντος, αλλά να επενδύσουμε στους καινοτόμους τομείς. Τώρα για την έκθεση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλής ποιότητος γιατί λαμβάνει υπόψη της τις δυσκολίες των περιφερειών που πλήττονται από την βιομηχανική κρίση. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε σήμερα στην Ευρώπη πώς θα καταφέρουμε να συνδέσουμε τη διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας με την επαναπεριφερειοποίησή της. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της έκθεσης λοιπόν είναι ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες και θα επιμείνω ιδιαίτερα τα εξής. Πρώτον, τη διαφάνεια των επιχορηγήσεων ιδιαίτερα στα κλώστερ και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως συμπεριλαμβάνονται και τομείς για τους οποίους δεν μιλάμε συχνά, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες, νέοι τομείς που έχουν αντισταθεί καλά στην κρίση και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ρόλο του πολιτισμού και της πολιτιστικής βιαμηχανίας για την καλύτερη εκμετάλλευση των πλητωμένων πρώην βιομηχανικών περιοχών. Μιλήσατε για τη Λίλη κυρία μου. Στη Λίλη υπάρχει ο σταθμός εμπορευμάτων του Αγίου Σωτήρος που έχει μετατραπεί σε καινούργια χρήση με ανακαίνιση των κτηρίων του και με ηλιακά. Επίσης μιλήσατε για νέα εργαλεία ολοκληρωμένης ανάπτυξης όπως τα IT. E Και αυτό είναι πολύ καλό για τον καθορισμό ολοκληρωμένων βιομηχανικών προγραμμάτων όσο κοντύτερα γίνεται στον πολίτη για να ανταποκρινόμαστε έτσι καλύτερα στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Επίσης όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα πολυπεριφερειακά προγράμματα όπου θα υπάρχει ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι βασικό για το μέλλον ότι χρειάζεται περισσότερη συνέργεια και συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου και των υπολείπων Ευρωπαϊκών Ταμείων, του Κοινωνικού Ταμείου μάλλον. Το Κοινωνικό Ταμείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόβλεψη και προσαρμογή στις ανάγκες των καινοτόμων τομέων, την επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και στην παιδεία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό για τομείς αναπτυσσόμενους, όπως τους πράσινους τομείς, δηλαδή τις, των ανεώσιμων πηγών ενεργείας, ας πούμε. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε πρότυπο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι τομείς αυτοί. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αντιποτελεσματικότερα το μέλλον. Ευχαριστώ. Η Μαρία Τερέζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την παρουσίαση και τις συγκεκριμένες προτάσεις που ακούστηκαν, ιδιαίτερα για την παράγραφο 5 που αναφέρει τις κύριες προκλήσεις. κρίση πλήττει κυρίως τις πρώην βιομηχανικές περιοχές. Στη Γαλλία υπάρχουν παραδείγματα όπως το Φλωράνζα ή η περίπτωση της Year και του Continental. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους καινούργιους άνεργους για τη μετεκπαίδευσή τους και τις επενδύσεις σε νέες υποδομές πιο ανταγωνιστικές και πιο αποτελεσματικές. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω, γιατί καμιά φορά ξεχνιέται, ότι το δημόσιο χρήμα δεν πρέπει τελικά να χρησιμοποιείται για τις μετεγκαταστάσεις σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην παράγραφο 6 ιδιαίτερα λέει ότι η Ευρώπη ξέχασε τις παλιές της βιομηχανικές περιοχές. Και επαναλαμβάνω όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα Θέλω να αναφέρω λοιπόν ιδιαίτερω την πρόταση που λέει και η μελέτη και η παρουσίαση να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τη στρατηγική της αναπροσαρμογής των πιο δημιουργικών τομέων που μπορούν να προσφέρουν και περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ανάπτυξη. Αυτού του είδους οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στις πρώην βιομηχανικές περιοχές. Όπως ας πούμε το παράρτημα του Λούβρου που άνοιξε στο Λάντς. Έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την τοπική βιοτεχνία, να επαναχρησιμοποιήσουμε τις πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως κινηματογράφους και θέατρα και έτσι να μετατραπεί η εικόνα ορισμένων πρώην βιομηχανικών πόλεων όπως η Γλασκόβη και η Λίλη σε κάτι άλλο. Δεν θα ήθελα να ξεχνάμε λοιπόν αυτήν την στρατηγική πολιτιστικής δημιουργίας που συχνά την ξεχνάμε στην απαρίθμηση βιομηχανιών. Ευχαριστώ Μαρή Τερέζ Λάμπερτ Βανιστερόι. Ευχαριστώ πολύ που συζητούμε αυτό το ζήτημα εδώ και το πραγματεύεται αυτό και η εκθέση και μελέτη. Καταρχήν να πω ότι αυτά τα τέσσερα παραδείγματα μας έδειξαν ότι η πολιτική συνοχή λειτουργεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και πρέπει να το λέμε. Γιατί αν δούμε τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και υπήρξε πραγματικά αλλαγή του τρόπου σκέψης σε σχέση με δύο-τρεις δεκαετίες πριν. Η ερώτηση μου είναι, ξέρουμε ποιες περιοχές ε, είναι υπό απειλή τώρα, ξέρουμε πού θα γίνει η επόμενη αναδημιουργία, που θα είναι η επόμενη σύγκρουση. Τώρα, στη δική μου περιφέρεια, δύο μεγάλες χημικές βιομηχανίες σταμάτησαν να λειτουργούν για διάφορους λόγους και αν δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, με την υψηλή τιμή της ε, ενέργειας σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ θα υπάρχουν μετακαταστάσεις όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς τις ΗΠΑ και προς άλλα μέρη του κόσμου. Ξέρουμε λοιπόν που να κοιτάξουμε που να ψάξουμε και έχουμε μια ευρωπαϊκή επισκόπηση για τους λόγους που μπορεί να επηρεάσουν τις εξέλιξεις τα επόμενα δέκα χρόνια. Στην αρχή είπατε κάτι. Ότι θέλετε να πείτε κάτι για την έξυπνη εξειδίκευση. Είπατε ότι μπορεί να αγγίξετε το θέμα κατά κάποιο τρόπο και κατόπιν αναφερθήκατε ε, στην ε, ε, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Όμως δεν πρέπει να δούμε μόνο την έρευνα και βιομηχανική ανάπτυξη. Υπάρχει τώρα στο πρόγραμμα Ορίζοντας. Έχουμε εκεί ένα κονδυλί 60-70 δισεκατομμυρίων διαθέσιμων και έχουμε και πολύ περισσότερα χρήματα μέσω των ταμείων ε, συνοχής. Αν ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, επομένω το συμπέρασμά σας θα μπορούσε να είναι ότι η πολιτική συνοχής ε, και το νέο που θετούμε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και τα δύο σημαντικό εργαλείο για την ανοικοδόμηση αλλά και για να εθετήσουμε νέες δραστηριότητες όπως είπε η Μαρή εγώ στη δική μου περιφέρεια είχα 10.000 ανέργους και τώρα έχουμε πολύ περισσότερο διαφοροποιημένη οικονομία με νέες εταιρείε που ε, διαδραστηριοποιούνται και στην τεχνολογία ε, όπως ε, βλέπουμε να είναι σημαντικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα συνδυασμό, να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη για να μπούμε στην εφάση. Και δεν βλέπω εδώ να υπάρχει αντίφαση. Μπορείτε να τοποθετηθείτε και εσείς σχετικά. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Λέω ο κύριος Φλάσακ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη αυτή σχετικά με τις ε, βιομηχανικές περιοχές, για όλα αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας δώσατε σε σχέση με την ε, μετατροπή των περιοχών αυτών. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη για μας. Θα ήθελα να τονίσω τα ακόλουθα. Αυτές οι περιοχές αποτελούν το 80% του ευρωπαϊκού επεπομένως πρέπει να προσδώσουμε την προσοχή μας σε αυτές. Και σήμερα μιλάμε πολύ για το θέμα της ανεργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση, το ITI. Εγώ θεωρώ ότι είναι το σωστό εργαλείο, το σωστό μέσο για αυτές τις ε, περιοχές. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Επομένως, το χαρτοφυλάκιο εγώ θα ήθελα να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, όπως με το πρόγραμμα Οριζόντας 2020 και αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ σημαντικό να διασυνδέσουμε με μονομένες στρατηγικές και πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου όταν δημιουργούμε αυτά τα προϊόντα δηλαδή διάφορες εθνικές, ευρωπαϊκές στρατηγικές, αλλά και τοπικές, αστικές ή περιφερειακές στρατηγικές. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες. Το leader ήταν μία από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν εδώ. Ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αστικές περιοχές. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το leader είναι κυρίως μία μέθοδος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα στις αγροτικές περιοχές, σε πιο μικρές περιοχές. Γιατί αν χρησιμοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει μία σύγκρουση μεταξύ των ε, τοπικών, ε, περιφερειακών, ε, αστικών αρχών, δημοτικών αρχών. Θα θέλαμε όμως εμείς να αποφύγουμε μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων εξουσιών. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια. Σας ευχαριστώ και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Χίμνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή ΕΝΒΗ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θέλω και εγώ να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία που συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το πρώτο σχόλιο Καταρχήν, ε, θέλω και εδώ να χαιρετήσω το ότι μπορούμε να συζητούμε τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για αυτή την διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά ποτέ δεν είχαμε λάβει υπόψη τη σημασία αυτής της στρατηγικής ε, για αυτές τις βιομηχανικές ε, ζώνες που λειτουργούν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις ε, παλιές βιομηχανικές ε, ζώνες. Μία καλή προστασία αυτών των περιοχών ε, θα επιτρέψει την ανθισή τους, την ανάπτυξή τους, όπως είπε και ο κ. Φενιστερόη, για να τις μετατρέψουμε με ένα φυσικό τρόπο, να τις συνοδεύσουμε στην ανάπτυξή τους και να δώσουμε κίνητρα για αυτή την ανάπτυξη προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία και μια πράσινη οικονομία, μιλώντας ευρύτερα. Δηλαδή, όχι μόνο να αναπτύξουμε πράσινους χώρους, αλλά να σκεφτόμαστε οικολογικά. Να υπάρχει έρευνα προσανατολισμένη στην οικολογία και έρευνα για την βιομηχανία, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε αυτές τις βιομηχανικές περιοχές ως ε, αποκλειστικά ένα μέσο παραγωγής, με πολύ πυκνό πληθυσμό, όμως η προσέγγιση αυτή δεν είναι η ορθή θα πρέπει να αντιληφθούμε διαφορετικά αυτές τις περιοχές και να τις δούμε ε, ως κάτι πολύπλοκο και να χρησιμοποιήσουμε και την έρευνα και την ανάπτυξη. Κάτι πολύ σημαντικό σήμερα είναι οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες αυτές οι βιομηχανικές περιοχές, οι παλιές βιομηχανικές περιοχές ε, μπορούν να, ε, να συμβάλλουν για μια ενεργειακή μετάλλαξη έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε όλη μας τη βαριά βιομηχανία. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε μια καμπή στην οικονομική ανάπτυξη Ήδη οι νέοι μας επλήττουν ότι δημιουργούμε αρκετές θέσεις εργασίας. Επομένως, αυτές οι περιοχές αποτελούν μια ευκαιρία αν τις αναπτύξουμε με έναν έξυπνο τρόπο. Αν η τοπική αυτοδίκηση καταλάβει ότι είναι ζωτικές αυτές οι περιοχές, ότι πρέπει να διατηρηθούν, Σίγουρα θα πρέπει να μετατραπούν, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εξαλειφθούν. Κάτι ακόμη. Αυτές οι βιομηχανικές λεκάνες βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές. Ε, σπάνιο είναι να έχουμε σιλικόν Valley όπως τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι περισσότερο ζώνες που βρίσκονται κοντά σε αστικές περιοχές ε, και διαφέρει η κατάσταση από ό,τι στην Αμερική. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε την καλή ανάπτυξη αυτών των βιομηχανικών τοποθεσιών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και ισορροπία σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές φορές, ε, όταν ε, βλέπουμε τέτοιες περιοχές ε, να εγκαταλείπονται, τότε εκεί διακόπτουμε και τις συγκοινωνίες. Όμως δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την επικοινωνία και μεταξύ αυτών των περιοχών και του υπόλοιπου αστικού ιστού. Θα πρέπει να μην φοβόμαστε να συνεργαστούμε με τους κατοίκους, ταυτόχρονα θα πρέπει και να τους εξηγήσουμε γιατί σχεδιάζονται οι τάδε δραστηριότητες στην τάδε περιοχή, ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό, μετατροπή της συγκεκριμένη ζώνης, αλλά σίγουρα να μην επιτρέψουμε την εγκατάλειψή της. Εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συζήτηση αυτή και εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και τις απόψεις σας και τα επιχειρήματά σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόεδρος, θέλει κάποιος... Κανείς να μιλήσει εκ μέρους της Κομισιόν. Όχι, ορίστε, ναι. Κύριε Κλάους Σούλτσε μου. Δεν προετοίμασα καμιά παρέμβαση, αλλά είδα τη μελέτη και τα συμπεράσματά της. Παρακολούθησα και τη συζήτηση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στην εξαιρετική ανάλυση που ακούστηκε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Γκάγερ για την εξαιρετική του έκθεση, μεταξύ άλλων και γιατί αναγνωρίζει ότι η δίκευση που προτείνεται εδώ μεταξύ περιοχών είναι πολύ καλό εργαλείο ανάπτυξης. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην κάνουμε ένα λάθος που συνήθως γίνεται, δηλαδή την μη πιστή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της Κομισιόν. η ειδίκευση μπορεί να παρεξηγηθεί ως αποκλισμός κάποιας περιοχής σε συγκεκριμένες μόνο δραστηριότητες, αλλά δεν εννοεί αυτό. Εννοεί με βάση τα στοιχεία που έχουμε των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων μιας περιοχής να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Δεν είναι μία εκ των προτέρων και από τα πάνω πρόταση που εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Και βέβαια εμείς από τα 11 θέματα που υποβάλαμε αυτά όλα περιορίζονται στο πρώτο. Είναι ένα μονοπάτι ώστε οι πρώην βιομηχανικές περιοχές να, μπορούν να, να μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση που τις πλήττει και να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες που έχουν και των ανθρώπων και του υπολείπου περιβάλλοντος. Και αυτό βέβαια απαιτεί και καλύτερο συντονισμό και κρατικά και με τα... το Περιφερειακό Ταμείο. Έχουμε διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και βλέπουμε πολύ θετικά θετικές πληροφορίες ως προς την ανταπόκρισή τους. Μερικές μάλιστα τώρα αρχίζουν να εφαρμόζουν τέτοια είδους καινούργια προγράμματα ενώ μέχρι τώρα δεν το σκέφτονταν καν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη στρατηγική μας. Έπειτα κάτι άλλο. Υπάρχει και το πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την περιφερειακή αυτή στρατηγική με μια γενικότερη πολιτική και εδώ ερχόμαστε στην περιφερειακή συνεργασία. τι θα γίνει με τα μελλοντικά προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας και πώς θα εκμεταλλευτούν καλύτερα τα κράτη-μέλη της ευκαιρίας που διαθέτουν ώστε να συντονιστούν και να εκμεταλλευτούν καλύτερα τους τομείς όπου μπορεί να εμφανίζουν κάποια αριστεία. Φυσικά αυτά συνδέονται και με τον λεγόμενο ορίζοντα 2020. Προετοιμάζουμε μια διάσκεψη για το θέμα και θα σας στηρίσουμε ενήμερους. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα τον κύριο και μετά την Κωνσταντσα. Την κυρία Τόντελινγκ δηλαδή. Ναι, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, αν ξέρουμε λέει ποιες περιφέρειες κινδυνεύουν λόγω της βιομηχανικής παρακμής. Η ανάλυση που έγινε για την πολιτική συνοχής βασίστηκε σε υποδομές και λοιπά. Εγώ δεν τα ξέρω βέβαια όλα, γιατί δεν είμαι παντογνώστρια για τη βιομηχανία. Νομίζω ότι δεν τα ξέρει κανείς όλα αλλά ίσως ο κύριος Σούλτσε από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο να γνωρίζει περισσότερα. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι είπε ότι η έρευνα δεν αντιφάσκει με όλα αυτά. Φυσικά δεν αντιφάσκει, αλλά φανταστείτε να υπάρχει μια περιφέρεια που προσπαθεί να προσαρμοστεί στις βιο... καινούργιες βιομηχανικές δυνατότητες δημιουργεί μία καινούργια πανεπιστημιούπολη ας πούμε. Πού θα ρίξει χρήματα η πολιτική συνοχή εκεί. Πού. Γιατί είναι καινούργιο και το ίδιο το θέμα και άρα δεν χρηματοδοτείται με τα παραδοσιακά κριτήρια. Εξαρτάται λοιπόν από την προοπτική του καθενός. Και ήθελα να πω ότι δεν γνωρίζουμε πολλά ως προς το πώς θα μπορούσε να δαπανίσει χρήματα η πολιτική συνοχή κάτω από τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα προγράμματα και κριτήρια. Στη Γενική Διεύθυνση Περίφ χαίρομαι που βλέπω τόσο μεγάλο ενθουσιασμό γιατί για τις περιφέρειες όπου γίνονται αξιολογήσεις εξάντε δεν είδα τόσο πολύ ενθουσιασμό για τα ΉΤΗ. ούτε διαπίστωσα στα γερμανικά ή αυστριακά κρατήδια να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τοπικές επενδύσεις δηλαδή για κονδύλια που να χορηγούνται από τα Υπουργεία. Δεν το έχω διαπιστώσει. Και η μέθοδος leader φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί για αστικές περιοχές. Ήθελα όμως να τονίσω ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου βρέθηκε μια μεθοδολογία και είναι λογικό να εφαρμοστεί μια προσαρμογή και τον ΙΤ e εκεί, όχι με την ίδια μέθοδο, γιατί 51% μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν μπορούν να αποφασίσουν για υποδομές, αλλά μπορούμε να συνδέσουμε και τα δύο θέματα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Δύο παρατηρήσεις. Εάν δεν ξέρουμε τι γίνεται σε μια, στη χημική βιομηχανία τα επόμενα δέκα χρόνια, ε, αυτό είναι τρομερό, διότι η επόμενη γενιά θα βρεθεί υπό ισχυρή πίεση παντού. Ίσως λοιπόν στην έκθεση Γκάιερ καλό θα, είμαι να, καλό θα είναι να είμαστε πιο προορατικοί. Και μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά, τα οποία ε, συχνά ε, ε συγκεντρώνονται σε κάποιες εταιρείες. Θα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επιπτώσεις. Και στις αστικές περιοχές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ολοκληρωμένο εδαφικό μέσο. Πρόκειται για επιλογή των τοπικών περιφερειακών και εθνικών αρχών το, το αν θα χρησιμοποιήσουν ε, αυτό το μέσο. Αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τις διάφορες πόλεις. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί. Είναι σημαντικό η αναδιάρθρωση τέτοιων περιοχών απαιτεί σημαντική αφοσίωση από πλευράς των κρατών μελών. Διότι θα πρέπει αυτή η πολιτική να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι θέμα απλά να βάλουμε τα χρήματα και να πούμε θα γίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Είναι θέμα εδαφικών παραγόντων, φυσικών παραγόντων. Σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με το θέμα των θέσεων απασχόλησης στο μέλλον, ε, να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση, διότι πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Ο κόσμος μερικές φορές πιστεύει ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν όσο έχουν, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε πολλά στην επόμενη γενιά και στους μελλοντικούς εργάτες. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε με, με ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά σημαντικό είναι να υπάρχει εθνική στρατηγική, η οποία να στηρίζεται από τις διάφορες πρωτεύουσες, να είναι διατεθειμένες ε, δηλαδή οι χώρες να επενδύσουν για τα επόμενα 10 χρόνια και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής να βοηθήσει το δικό μας ε, εδαφικό μέσο, ε, αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη να επιφέρει αυτή την αλλαγή. Καλά, μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες Νομίζω ότι τα θέματα αυτά θα είναι ακόμη πιο σημαντικά τα επόμενα δέκα χρόνια. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαι υπερβολικά γενναιόδορη με το χρόνο ομιλία που δίνω. Πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ε, τη, η μόνη απόφαση που πρέπει να λάβουμε αυτή τη στιγμή είναι να θέσουμε την προθεσμία για τις τοπολογίες που είναι 21 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τρέτλινγκ. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο θέμα 5 της ημερησίας διάταξης. Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη, μια οικονομία για την Ευρώπη και δίνω το λόγο στη Ρίκα Μάνερ για να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Καταρχήν αυτή η βιοοικονομία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, τομέας ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Από τη σκοπιά της περιφερειακής ανάπτυξης επίσης ε, στο μέλλον αυτή η βιοοικονομία παρουσιάζει πολλές δυνατότητες για την Ευρώπη και πηγή απασχόλησης. Η βιοοικονομία αποτελεί μια ευφυή, e, μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία, κυρίως στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020. Τώρα, από τη σκοπιά της περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να σκύψουμε στα διάφορα θέματα που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία και θα πρέπει να σκύψουμε σε αυτή την ευφυή e οικονομία, γιατί εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο για να καταρτήσουμε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όπως είπα, πολλά πρέπει να βελτιωθούν, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες επίσης. Θα πρέπει να πράξουμε έτσι ώστε η οικονομία να παράγει ευφυή προϊόντα σε ό,τι αφορά την αηφορία και την ανάπτυξη. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και τον έξυπνο τρόπο χρήσης αυτών των πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα όσα αφορούν ε, τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας και επίσης θα πρέπει να μιλάμε και για εξειδίκευση. Σήμερα αυτή η βιοοικονομία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τα νέα υλικά, για τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα κτλ. Εδώ μιλάμε για τομείς ανάπτυξης για το μέλλον και για τομείς μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων θα έπρεπε να επικεντρώσουμε τις πηγές μας, τους πόρους, συγγνώμη, σε αυτούς τους τομείς, κυρίως όταν μιλάμε και για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους στη δασοκομεία. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής θα πρέπει να επιμείνουμε στα στοιχεία και τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε το δυναμικό μας σε, περιφερειακή, σε περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα. Στο πλαίσιο αυτό θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό και περισσότερη χρηματοδότηση. Επίσης, να μην ξεχνάμε πως ε, όταν στρεφόμαστε προς τη βιοοικονομία, χρειαζόμαστε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Ε, επίσης, πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μία νομοθεσία σαφή, για να αναπτύξουμε τους απαραίτητους πόρους, την απαραίτητη χρηματοδότηση για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να έχουμε και την απαιτούμενη ανάπτυξη. Όπως σας είπα, η βιοοικονομία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για αυτή την ευφυή ανάπτυξη και επιμένω στο ότι οι περιφέρειες έχουν αυτή τη γνώση στη διάθεσή τους για να θέσουν σε εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Οι περιφέρειες μπορούν να ενεργοποιήσουν ε, τα διάφορα είδη βούλησης. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε να υπάρχει ενεργοποίηση σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καθολική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα διάφορες εξειδικεύσεις, στους διάφορους τομείς. Χρειαζόμαστε προγράμματα, ε, δημόσιες ιδιωτικές συμπράξεις, συμπράξεις ιδιωτικού δικαίου και είναι πολύ σημαντικό οι μικρές και μισές επιχειρήσεις ε, να τεθούν σε πρώτο πλάνο. Γιατί Αυτές αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μπορούν να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση αυτή. Επιπρόσθετα, σε αυτή τη γνωμοδότηση επιμένω στο πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση σε περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους σε περιφερειακό επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να επιμένουμε να υπάρχει κατάρτιση και εδώ έχω κατά νου και την ε, εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση. Για να ολοκληρώσω, επιμένω και πάλι στο ότι θα πρέπει να θέσουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά παντού στην Ευρώπη. Αυτή η βιοοικονομία θα ήταν καλό να τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Τώρα να περάσουμε στους κοιόδες. Λαμπέρ για το ΕΛΚ. Πολύ σύντομα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρίκα Μάνερ που με πολύ σωστό τρόπο αναφέρεται στην πτυχή της ε, περιφερειακής πολιτικής. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά θα ήθελα πρώτα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είναι πρώτη φορά που η Κομισιόν υποβάλλει μια ολοκληρωμένη θέση για τη βιοοικονομία. Παλαιότερα είχαμε λίγα πράγματα εδώ, λίγα πράγματα εκεί, Λίγα για την ε, γεωργία, λίγα για την έρευνα και ανάπτυξη, λίγα για τη βιομηχανία, αλλά τώρα έχουμε κάτι για έναν ενιαίο τομέα. Και είναι ε, πολύ χρήσιμο το ότι γίνεται η σύνδεση με την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Θέλουμε λοιπόν ε, θέσεις απασχόλησης πιο ευφυείς και πιο πράσινες. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε προσπάθειες για τα θέματα αυτά. Και μπορούμε να συμβάλλουμε ε, στα προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, κλπ. Θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες ε, και είμαι περίεργος ε, να δω ποια είναι τα εμπόδια για την έξυπνη εξειδίκευση, την ευφυή εξειδίκευση και σε, ποιους, σε ποιες περιφέρειες θέλουμε να δούμε την τη σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, προϊόντα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από ε, νέα υλικά ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα όσα λέει η συντάκτρια. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε την, ε, τις δυνατότητες συνέργειας που υπάρχουν και για την επόμενη 7 ετία έχουμε βασιστεί σε νέα υλικά. Είναι πολύ καλό το ε, να συνδέσουμε τις ε, πτυχές αυτές ε, με τα όσα γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο για, με τα ΚΙΚΣ, ε, ε, με τα, κέντρα καινοτομία. Ε, να εξετάσουμε το θέμα αυτό, μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία για κάποια θέματα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για τη δουλειά της. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή που τη βρίσκω λογική μπροστά στις πιέσεις που αντιμετωπίζουμε για το περιβάλλον και την υπερεκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων. Πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει μία νέα αντιμετώπιση και παραγωγής και κατανάλωσης, βιώσιμη και μόνιμη. Η βιοοικονομική στρατηγική μας φαίνεται καλή βάση για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτά τα προβλήματα για μια κοινωνία που θέλουμε να είναι πιο ανταγωνιστική και λιγότερο ακριβή. Θα ήθελα να επιμείνω ότι η βιοοικονομία είναι μια πραγματική ευκαιρία για ανάπτυξη στις περιφέρειές μας εφόσον διαθέτουν βέβαια τις δεξιότητες, τις απαραίτητες δεξιότητες, αλλά δεν αρκεί. Η συγκέντρωση της προσοχής στην έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να είναι βασική και να υπάρξουν επενδύσεις στις περισσότερες δεξιότητες και γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο ένα πιο λογικό πολιτικό πλαίσιο αλλά και επένδυση σε νέες υποδομές και σε δημιουργία νέων εργαλείων και κριτηρίων πανενωσιακός. Θα ήθελα να επιμείνω στη σημασία που έχει κινητοποίηση των πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το περιβάλλον και η βιοοικονομία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν συμβάλλει σε αυτό αν δεν συμβάλλουν σε αυτό και οι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να έχουν καλή πληροφόρηση για να αναπτυχθούν και τοπικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες. Είναι εξάλλου ένας από τους στόχους της δημοσίευσης της Κομισιόν αυτός στον πρακτικό οδηγό για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. Και για μένα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όπως και η κυρία Μάνερ τον αποφασιστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οποίες πρέπει να εγγυηθούμε δυνατότητες χρηματοδότησης. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες για την έρευνα, τη χρησιμοποίηση νέων εργαλείων χρηματοδότησης και καλύτερης δικτύωσης και διάδοσης των πληροφοριών και γνώσεων. λέει και η εισηγήτρια πρέπει και περιφερειακά να εγγυηθούμε μια επαγγελματική, τεχνική και γενικότερη εκπαίδευση που να στοχεύει σε υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία. Τέλος, Επιμένω να παρακολουθήσουμε και με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη όλων αυτών και χαιρετίζω εδώ την πρωτοβουλία της Κομισιόν να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο της βιοοικονομίας και μια επιτροπή εμπειροχνομόνων. Να υπάρχει δηλαδή σαφές πρόγραμμα και οδικός χάρτης. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Χρυσόγελος. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την συγγήτρια γιατί είναι ένα θέμα που σχετίζεται και με την προηγούμενη κουβέντα νομίζω για το θέμα της ε, βιομηχανικής πολιτικής. Γιατί πρόκειται για μια μεταστροφή πραγματικά ενός ολόκληρου κύματος βιομηχανίας που γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες σε ένα άλλο μοντέλο βιομηχανίας το οποίο βασίζεται πολύ στην αποκέντρωση, βασίζεται πολύ σε πρώτες ύλες που είναι αποκεντρωμένες περιφερειακά και βασικά πρέπει να βασίζεται και σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Άρα πράγματι έχουμε μια αναδιάρθρωση της βιομηχανίας όπως την ξέραμε, αν ακολουθήσουμε το μοντέλο της βιοοικονομίας και αυτό πρέπει να γίνει βέβαια με ένα βιώσιμο τρόπο για να αποφευχθούν προβλήματα ή κίνδυνοι, γιατί από μόνη της η βιοοικονομία δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ε, μηδενικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύχθηκε η παραγωγή βιοκαυσίμων σε βάρος της παραγωγής τροφίμων, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε πιθανούς κινδύνους που έχουν σχέση με την απώλεια βιοπικιλότητας, με την ε, κακή διαχείριση των δατικών πόρων ή συγκρούσεις προτεραιοτήτων και αναγκών, π.χ. μεταξύ παραγωγής τροφίμων και παραγωγής καυσίμων, βιοκαυσίμων για οχήματα. Αυτό μας ε, οδηγεί νομίζω και σε μια συζήτηση για το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με την ε, βιοοικονομία. Πάντως όμως η βιοοικονομία είναι ένα κλειδί για να πετύχουμε στόχους όπως είναι η οικονομική, κοινωνική και ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συνδέεται απόλυτα με περιφερειακές πολιτικές και δίνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα στις περιφέρειες να αναπτύξουν ένα δικό τους μοντέλο οικονομίας, περιφερειακά οργανωμένης, το οποίο δεν είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συχνά, βασισμένες σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ορυκτά καύσιμα. Άρα λοιπόν η βιοοικονομία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και μπορεί να αποφεληθεί εφόσον υπάρχουν συγκροτημένες σε κάθε περιφέρεια στρατηγικές για την ανάπτυξη οικονομίας με βάση τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά ε, από άψη περιβάλλοντος, από γνώσεων, τεχνοσίας, ε, ανανεώσιμων ε, ε, πόρων και πρώτων υλών που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της βιοοικονομίας. Για παράδειγμα, Πολλέ περιοχές δεν έχουν δικό τους πετρέλαιο, δεν έχουν δικό τους φυσικό αέριο, πρέπει να το εισάγουν. Όμως πολλές αγροτικές περιοχές θα μπορούσαν να αξιοποιούν τα υπολείμματα γεωργικής δραστηριότητας ή τα υπολείμματα από τη διαχείριση δασών, κάτι που ήδη έχουν κάνει αρκετές ε, περιοχές στην Ευρώπη και άρα μπορούν να, έχουν, να απεξαρτηθούν ή να μειώσουν τουλάχιστον την εξάρτησή του από εισαγόμενα ε, ορυκτά καύσιμα ή γενικότερα από εισαγόμενες ε, πηγές ενέργειας. Ε, πρέπει βέβαια να υπάρξει πραγματικά ένας διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και τώρα που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως η στρατηγική για την ε, βιοοικονομία, να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση σε πολλές περιοχές, γιατί πολλά από αυτά που ε, συζητάμε για βιοοικονομία υπάρχουν εδώ και αιώνε. Η παραγωγή του τυριού ή του κρασιού ή τη μπύρα είναι μορφέ βιοοικονομία. Η παραγωγή βέβαια βιοπλαστικών είναι κάτι άλλο. Είναι μια, βασίζεται σε σύγχρονε έρευνε. Αλλά μπορούμε αξιοποιώντα και την παράδοση περιοχών και τι έρευνε και τι γνώσει επιστήμη να διαμορφωθούν σε κάθε περιφέρεια οι στρατηγικέ για την ε, βιοοικονομία. Ε, υπάρχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι οι μορφές βιοοικονομίας μπορούν να στηριχθούν ε, κατά βάση σε μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει και συνεταιρισμού. Και εδώ αλλάζει και το μοντέλο τη βιομηχανία συνολικά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έχουμε μια βαριά βιομηχανία και τεράστιε ε, βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και στην πιο μικρή περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία που έχει χαρακτήρα και ε, πράσινης βιομηχανίας και έτσι να υπάρχουν συμπληρωματικέ θέσει εργασία και να συμπληρωθεί ο αγροτικό τομέα, παράδειγμα, με μοντέλα παραγωγής ενέργειας που βασίζονται στη βιοοικονομία. Άρα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Για να πετύχουμε όμως αυτές τις αλλαγές, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη αναδιάρθρωση της οικονομίας, χρειάζονται και στοχευμένες παρεμβάσεις στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην ε, Κοινωνική Συνοχή. Αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ε, ενισχύσουν αυτές τις, τη μεταστροφή αυτή προς την ε, ε, βιοοικονομία. Και τέλος θα ήθελα να κλείσω να πω ότι υπάρχει μόνο ένας σοβαρός κίνδυνος τον οποίο θα πρέπει τουλάχιστον εμείς οι πράσινοι θεωρούμε ότι πρέπει να αποκλειστεί. Είναι στο όνομα της βιοοικονομίας να στραφούμε στα γενετικά, τροποποιημένα, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στη λογική ότι θα κάνουμε έτσι πιο αποδοτική την βιοοικονομία νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούμε στη γενετική ποικιλότητα και στην ποικιλομορφία που υπάρχει, γιατί μπορεί και η βιοοικονομία να οδηγηθεί σε μια πλήρη εξάρτηση από ορισμένες επιχειρήσεις. Και βέβαια να έχουμε και άλλα σοβαρότερα προβλήματα μετά στο περιβάλλον από την υπερβολική χρήση ε, οργανισμών που έχουν φτιαχτεί στα εργαστήρια. Ευχαριστώ κύριε Σουλασάκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η βιοοικονομία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη γιατί προστατεύει τις μη ανανεώσιμες πηγές και προστατεύει και τις ανανεώσιμες πηγές. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος το Φεβρουάριο η Κομισιόν δημοσίευσε μια στρατηγική σχετικά με τη βιοοικονομία και αναφέρεται και στο παρατηρητήριο που θα ιδρύθει φέτος και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της βιοοικονομίας. Και επειδή είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, μόνο πέντε κράτη-μέλη έχουν μία στρατηγική βιοοικονομία Φιλανδία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία και κάτω χώρες αν ε, πρόκειται να προβούμε σε συντονισμό, θα πρέπει να πούμε τι πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπε χώρες ε, και πώς ε, από κοινού θα παρουσιάσουν κάποια σχέδια. Επίσης, το παρατηρητήριο αυτό θα έχει το δικό του προπολογισμό και το δικό του προσωπικό και θα ήθελα να ξέρω πώς η Κομισιόν θεωρεί ότι θα λειτουργήσει αυτό το παρατηρητήριο από αυτή τη σκοπιά. Κομισιόν, θέλετε το λόγο. Δεν έχουμε κάποιο όνομα από την Κομισιόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπο, Παρακαλώ. Μπορείτε να μας πείτε και πώς λέγεστε. είμαι Σίλβια Νέιμαντ από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, από την Αρμόδια Διεύθυνση ε, για την ανακοίνωση, που δημοσίευσε την ανακοίνωση. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και την Συγγήτρια για αυτή την εξαιρετική γνωμοδότηση και θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα σημεία που τέθηκαν από τους κλειώδεις συζητητές η Κομισιόν γνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της στρατηγικής για την οικονομία και το σχεδίου δράσης εξαρτώνται από το πώς θα εφαρμοστούν αυτά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε στενά με τους περιφερειακούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ε, δημοσίευσε και μία γνωμοδότηση στο τέλος του περασμένου έτους για τη βιοοικονομία και τόνισε και το ρόλο ε, της εφαρμογής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, αναγνωρίσαμε την ανάγκη να οικοδομήσουμε συνέργειες μεταξύ των διαθετικών ταμείων και του ορίζοντα 2020, της κοινή γεωργικής πολιτικής, ακόμη και της κοινή ελευτικής πολιτικής. Επομένως, τα γνωρίζουμε όλα αυτά και παίρνουμε το χάρη τον οδηγό για την ε, FEE εξειδίκευση που παρουσίασε η ΓΔ Ρίτζο για τις ε, τοπικές αρχές τονίζεται ότι πολλές από τις επενδύσεις που έχουν ε, ήδη λάβει χώρα έχουν σχεδιαστεί να ενταχθούν στις στρατηγικές τους θα πρέπει να εμπίπτουν στην πολιτική για τη βιοοικονομία. Επομένω, αυτό εξαρτάται τελικά από τα κράτη-μέλη αν θα το επιλέξουν, αλλά εμεί ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί επιπρόσθετα να υπογραμμίσω την πτυχή της ευαισθησία των καταναλωτών ε, για όλες τις ψυχές της βιοοικονομίας. Μιλήσαμε πολύ για το γενικό ρόλο της εκπαίδευσης, της παιδείας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε να εμπλέξουμε και τις νέες γενιές στους τομείς της βιοοικονομίας. Παρ' όλα αυτά, Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των πληροφοριών στους καταναλωτές και πώς θα κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, δηλαδή να αγοράζουν και τέτοια προϊόντα που βασίζονται στη βιοοικονομία και να δημιουργηθεί και μία ΣΔΙΤ ε, για αυτά τα προϊόντα που βασίζονται στην οικονομία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διατομεακή και μεταξύ όλων των επιπέδων, περιφερειακού, εθνικού, ευρωπαϊκού επίπεδου. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ε, εκπόνηση εθνικών στρατηγικών βιοοικονομίας, είναι αλήθεια ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι πιο προχωρημένα. Παρ' όλα αυτά, Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και την εκπόνηση τέτοιων στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί μπορεί να είναι σημαντικό για να συνδυαστούν διάφορες ναι. και σε ό,τι αφορά το παρατηρητήριο που πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί, ο στόχος θα είναι να αξιολογεί τακτικά τον αντίκτυπο της βιοοικονομίας και την πρόοδο της και μπορεί να συμβάλλει στην εκπόνηση αυτών των ε, στρατηγικών βιοοικονομίας στο παρατηρητήριο. Ε, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει να λειτουργήσει συνεργασία με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, το JRC, και περιμένουμε αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω εφαρμογή της στρατηγικής βιοοικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μίλησε. Πολύ σύντομα. Άκουσα αυτά που υπόθηκαν και αναρωτιέμαι. Μιλήσατε για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την σημασία της σύνδεσης ανάμεσα στη βιοοικονομία και στη κοινωνική οικονομία, διότι και η κοινωνική οικονομία είναι πολύ σημαντική. Η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων για να λύσουν τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή τη σχέση. Ρίκα θέλεις να σχολιάσεις. Ναι, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα ωραία τους σχόλια. Ελπίζω να μεταφραστούν όλα αυτά και σε συγκεκριμένες τροπολογίες. Όπως υπόθηκε πολλές φορές, Εδώ μιλάμε για ουσιώδη πράγματα που πρέπει να τα λέμε πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρη σειρά υλικών που πρέπει να τα αναπτύξουμε για να έχουμε μια βάση βιοοικονομίας. Δηλαδή, έχουμε γνώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι κάτι το βασικό. Ας μην τις έλθω σε λεπτομέρειες, όλο, να σχολιάσω όλα όσα ακούστηκαν, γιατί γενικά οι παρατηρήσεις ήταν ενδιαφέρουσες και ελπίζω να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 22 Μαρτίου το μεσημέρι. Και τώρα το επόμενο σημείο το 6. Προγραμματισμός πολιτικής και με τάσεις δύο τελείες δημοσιονομικές επιπτώσεις δημιουργίας ικανοτήτων τελεία. Ο κύριος Βλάσακ. Κυρίες και κύριοι, σας κατευχαριστώ. Ο προβλεπόμενος σχεδιασμός είναι κάτι βασικό για τους προϋπολογισμούς μας όλων. Με βάση την επικουρικότητα είναι σαφές ότι οι μακροπρόθεσμες κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές και προγράμματα καθορίζουν μέσω διαφόρων αρχών και οργανισμών το συντονισμό, τον προϋπολογισμό. Για να ενδυναμώσουμε δε τον εξυγχρονισμό της διοίκησής μας πρέπει να έχουμε ορισμένους πόρους για το σχεδιασμό. Έχουμε το κοινωνικό ταμείο και το περιφερειακό ταμείο βέβαια. Τα έχουμε αυτά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ΜΗΣ όπως την καταπολέμηση της διαφθοράς ή τη μείωση του διοικητικού άχθους των επιχειρήσεων ή για τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης ανθρωπίνων και άλλων πόρων στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικό να σχεδιαστεί όπως πρέπει, επειδή ακριβώς είναι πολιετές. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ του εθνικού και του ενωσιακού επίπεδων. Όταν διατυπώνουμε προτάσεις για πολιτική, ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες τάσεις που παρατηρούνται Χρειάζονται λοιπόν μελέτες ε, που έχουν ήδη παραγγελθεί και προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ευρώπη 2030 η μελέτη Ευρώπη 2030 που έγινε από το Συμβούλιο ή ανάλογη μελέτη από άλλες ανάλογες μελέτες από άλλες υπηρεσίες της Ένωσης. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των τάσεων. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο συντονισμό και συνεργασία ώστε να καταλήξουμε σε ένα διαθεσμικό σύστημα που να είναι σε θέση να ταυτίζει τις τάσεις και να συμπεριλαμβάνει όλους τους παράγοντες και μεταβλητές με καλύτερη χρησιμοποίηση και του προσωπικού όλων, όλων των ευρωπαϊκών θεσμών μεταξύ των οποίων και την Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτά είχα να σας πω και προσβλέπω στα σχόλια και παρατηρήσεις σας. Μόνο ο Αλφόνση νομίζω είναι από τους Κιώδης, επομένως θα πάρει αυτό το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί για τα ταμεία συνοχής νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για να βοηθήσουμε τους διάφορους πρωταγωνιστές ε, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, των ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Είναι κρίμα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε μια τέτοια συνήθεια. Ίσως θα μας επιτρέψει αυτή η έκθεση να ξεκινήσουμε σε κάτι τέτοιο δηλαδή, στο να έχουμε ένα καθολικό σκεπτικό και να εμπλέκουμε και τις περιφέρειες για να λάβουμε υπόψη και τις ε, τοπικές ανάγκες αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει και η για τους προσανατολισμούς που θα πρέπει να αναλυθούν ε, κτλ. Εγώ λοιπόν φυσικά είμαι υπέρ όλων αυτών των ζητημάτων και νομίζω ότι οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε ε, μπορεί να είναι χρήσιμες κυρίως ό,τι αφορά το θέμα της εφαρμογής ε, της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ, Λαμπέρ Φανιστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάπως δύσκολο να καθορίσουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται εδώ. Συζήτηση ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχετικά με περιοχές, πολιτικές, με περικοπές, συγγνώμη, ε, πολιτικές λιτότητας. Το θέμα της δημιουργίας ικανοτήτων, λοιπόν, και της διασφάλισης σε όλα τα επίπεδα επαρκούς εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ε, είναι σημαντικό ε, όταν κάποιος ε, κρατάει στο, χέρι τα χρήματά του, όλοι ζητάνε περικοπές, αν όχι όλοι θέλουν αύξηση ικανοτήτων. Ε, στα σημεία 6 και 7 ιδιαίτερα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπως ε, πιο ανοιχτή απέναντι στα όσα έχουν ε, επιτευχθεί. Είναι σημαντικό το θέμα της επικουρικότητας στα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ε, ίσως ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς έχουμε κάνει τα πράγματα μέχρι τώρα ε, και να προχωρήσουμε και στο naming and shaming, τον κατονομασμό των ενόχων. Ας κοιτάξουμε την Ισπανία. Τι πρέπει να γίνει για να δημιουργήσουμε εκεί τις απαραίτητες ικανότητες και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Διότι εάν ε, κάποιος ε, ήδη ε, βρίσκεται στην αγορά εργασίας μπορεί να έχει καλύτερες ελπίδες από κάποιον που τώρα μπαίνει στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το θέμα των δεξιοτήτων, των επενδύσεων στους διάφορους τομείς. Θα πρέπει όμως να δούμε και επικριτικά την πολιτική υπό τη μορφή που έχει σήμερα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει. και σίγουρα μπορούμε να συμβάλλουμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, δεν είμαι βέβαιος αν είναι ακριβώς αυτό που ζητάει ο Βλασάκ. I don't see anybody Ευχαριστώ. πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο ε, το λόγο. Θα παρακαλούσα λοιπόν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να πάρει το λόγο. Έχουμε ε, εδώ τον ε, Πάσκο Κάλ από το γραφείο του κυρίου Παρόσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το λόγο θα πάρει ο συνάδελφός μου, Κρέιαμ, που θα παρουσιάσει ε, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην Επιτροπή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μου δίνει τη δυνατότητα αυτή να πω λίγα λόγια σχετικά με ε, ένα από τα προγράμματα ε, δημιουργίας ικανοτήτων που ε, εξετάζουμε σε όλα τα θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Χρειάζεται λοιπόν μια στρατηγική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις πολιτικές που έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό με τον ίδιο τρόπο που εξετάζεται και αλλού, στη Washington, ε, στο Δελχή και στη ε, στην Beijing. Έχουμε λοιπόν ε, το ΕΣΠΑ σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 2010-2011 και η Ένωση ξεκίνησε έτσι μια διαδικασία με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και, την, και να βοηθήσει ε, ε, όσο ασκούν πολιτική στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με βάση εμπειρικά στοιχεία και προορατικότητα. Το πιλωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012. Είχαμε μια έκθεση που λεγόταν «Παγκόσμια στάση το 2030». Στην έκθεση αυτή αναφέρθηκαν διάφορες στάσεις οι οποίες θα διαμορφώσουν τον κόσμο το 2030 που είχε να κάνει με την αποσχολησιμότητα του ατόμου, την ε, αύξηση των δυνατοτήτων, ε, την ε, δημιουργία ενός πολυκεντρικού κόσμου και τέλος τα διάφορα κενά ε, στη διακυβέρνηση που θα πρέπει να καλυφθούν. Η πρόοδο στο πολιτικό αυτό πρόγραμμα επέτρεψε στην ΕΣΠΑΣ να προχωρήσει σε μια δεύτερη ε, φάση με δεύτερη γραμμή του προπολογισμού που συμφωνήθηκε στο προπολογισμό του 2012. Η δεύτερη φάση από το 2012 μέχρι το 2013 καλύπτει τρεις βασικούς τομείς αναλύσεων. Πρώτον την οικονομία, δεύτερον κοινωνικές αλλαγές και τρίτον διεθνής διακυβέρνηση και εξουσία. Οι τρεις μελέτες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή θα ε, δείξουν βασικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και το χρονοδιάγραμμα μας ε, επικεντρώνονται στο 2030. Στόχο έχει να προβλέψει προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κύκλο πολιτικής 2014-2019. Η διαθεσμική ομάδα που εξετάζει το θέμα αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και εξετάζει ιδιαίτερα τα οριζόντια θέματα στην οικονομία, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η εφαρμογή των τριών μελετών που έχει προγραμματιστεί για τον φετινό Σεπτέμβριο πραγματοποιείται υπό την εποπτεία μιας διαθεσμικής ομάδας και τριών ε, ειδικών ομάδων ε, όπου συμμετέχουν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι σχετικές μελέτες θα αποτελέσουν την αναλυτική βάση για την προετοιμασία ε, της Διευθύνουσας Ομάδας της ΕΣΠΑΣ θα εκπονηθεί λοιπόν μια έκθεση με βάση τις τρεις μελέτες ε, που ανέφερα και θα εντοπιστούν οι διασυνδέσεις ε, και θα καθοριστούν τα βασικά θέματα για την ευρωπαϊκή πολιτική για τον επόμενο κύκλο και μετά από αυτόν και η τελική έκθεση προβλέπεται να είναι διαθέσιμη αρχές του 2014. Ελπίζουμε εγκαίρως για τις ε, μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν σε διαθεσμικό επίπεδο εντός ε, του 2014. Έτσι λοιπόν ελπίζω να σας έχω δώσει μια ευρία επισκόπηση του προγράμματος, ε, αλλά... Για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο εισηγητής και οι σκιώδει είναι ότι αυτό που γίνεται στην ΕΣΠΑΣ είναι μια σαφή απάντηση σε μια σαφή ε, ανάγκη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, αλλά σε διαθεσμικό επίπεδο και όχι μόνο εντός του κάθε θεσμικού οργάνου. Ε, εγώ συμμετέχω σε μία από τις ομάδες εργασίες και εξετάζω και βλέπω την σχέση μεταξύ του προσωπικού των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ε, εδώ ε, μια, ένα νέο επίπεδο δημιουργικότητας και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το σύστημα μόνιμο, να υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα Ε, πώς θα γίνει η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων ε, των εργασιών της ΕΣΠΑΣ, ε, τι περιμένετε από το Κοινοβούλιο και... και στα άλλα θεσμικά όργανα. Ε, οι διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις ε, της Κομισιόν θα μας πούνε για την εφαρμογή των συστάσεων. Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι, Πρόεδρε. Ε, όπως είπε ο συνάδελφος, πρόκειται για το μόνο διαθεσμικό πρόγραμμα που έχουμε, το οποίο σημαίνει ότι η διευθύνουσα ομάδα που επιβλέπει το πρόγραμμα ε, αποτελείται από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν. Και η ομάδα αυτή θα βασιστεί στα συμπεράσματα των διαφόρων εκθέσεων που θα πρέπει να προετοιμαστούν από τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και θα υποβάλουν μια οριστική έκθεση αρχές του 2014 με τις πολιτικές συστάσεις. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε επίπεδο ομάδων εργασία. Υπάρχουν τρεις ομάδες ε, μία για την οικονομία, μία για κοινωνικά θέματα και μία για τη διακυβέρνηση. Εγώ προεδρεύω της ομάδας ε, για την οικονομία και ε, το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά όπως ε, και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φα... Στη δεύτερη φάση η διευθύνουσα ομάδα θα εκπονήσει η έκθεση η οποία θα σταλεί στα θεσμικά όργανα στις αρχές του 2014. Οι συστάσεις λοιπόν των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου θα εξεταστούν από την ε, Κομισιόν και θα εφαρμοστούν από την Κομισιόν και το ε, Κοινοβούλιο στις διάφορες ε, ομάδες εργασίας. Εξέτασα το σχέδιο του εισηγητή, το οποίο ταιριάζει πολύ καλά με τις προθέσεις της Κομισιόν για τα επόμενα χρόνια. Thank Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα από αυτού και αν θα μπορούσατε να σκεφτείτε δύο φορές επί των συστάσεων για το τι θα θέλατε να δείτε για την πραγματική λειτουργία όλης αυτής της διαδικασίας. Έτσι ώστε η πολιτική συνοχή, η περιφερειακή πολιτική είναι η κύρια επενδυτική πολιτική και να μην παραγκονιστεί. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που λάβουμε αυτές τις πληροφορίες σήμερα και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί και η έκθεση. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια, να ξαναρωτήσω τον συγχητή αν θέλει να κάνει κάποιο τελευταίο σχόλιο. Όχι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τις πληροφορίες, θα είμαστε επικοινωνία για να αποσαφηνίσουμε κάποια ζητήματα, για να κάνω κάποιες αλλαγές στην εκθεσή μου και επίσης ε, θα ήθελα θα έρθω και σε επικοινωνία με τον αρμόδιο της Επιτροπής Προπολογισμών. Ευχαριστώ προς το παρόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακόμα πότε θα είναι η τελική ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή, αλλά οι τροπολογίε πρέπει να κατευθούν ε, μέχρι τις 22 Μαρτίου για την τελική ψηφοφορία στη τέλη Απριλίου, στην περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή θα ψηφίσει το Μάιο. Προτείνω λοιπόν 22 Μαρτίου το μεσημέρι ως καταλεκτική ημερομηνία να κλείσουμε αυτό το σημείο τώρα στη μερική διάταξη. Σας ευχαριστώ κομπισιόν. Λοιπόν, και όσον είναι εδώ. Έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας, αυτό είναι καλό για ένα ευρωπαϊκό όργανο. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της γαλλική ανάπτυξης, πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλασσιών μεταφορών και του τουρισμού. Παρακαλώ. Σόν, από είσαι έτοιμος, ναι είμαι έτοιμος, ευχαριστώ πολύ. Εσείς ε, πάντοτε είστε μπροστά στο χρόνο, μην ανησυχείτε, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχω αναλάβει αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι το έγγραφο της Κομισιόν μας ε, παρουσίασε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα πραγματικής ανάπτυξης και δημιουργίας ε, θέσεων εργασίας και βιωσιμότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βέβαια θα έχουμε τη σωστή υποδομή. Και αυτή θα είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί καταρχήν χρειαζόμαστε υποδομές για την ανάπτυξη του δυναμικού της θάλασσας. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ασφαλεία δικαίου και επίσης και εμπιστοσύνη για όσους θέλουν να επενδύσουν ε, σε πολλούς από τους ε, τομείς, όπου υπάρχει αυτό το τεράστιο δυναμικό ως προς την ανάπτυξη. Και εγώ παρουσιάζω ορισμένου από τους τομείς εδώ, που νομίζω ότι είναι πολυπρακτικού χαρακτήρα και φυσικά το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για εθνικού ε, πόρου και για εγχωρία υδάτα. Αυτό σημαίνει ότι εδώ μπαίνει ο κεντρικό ρόλο τη Επιτροπή μα, γιατί τα θαλάσσια ζητήματα είναι θέματα ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε αυτέ τι προτάσει. Νομίζω ότι οι αποτελεσματικοί πόροι πρέπει να στοχοθετηθούν, θα πρέπει να υπάρχει streamlining έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές αυτές θα έχουν έναν ορθό αντίκτυπο για την ε, ανάπτυξη. Στο σχέδιο της γνωμοδότησής μου, εγώ καλώ να επικεντρωθούμε στις συνέργειες μεταξύ των διάφορων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε τα ναυτιλιακά κλάστερ και ορισμένες ε, πρωτοβουλίες υπάρχουν ήδη σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει και το πρόγραμμα της δική μου χώρα, το Infomar, το οποίο δίνεται εδώ ως παράδειγμα στο κείμενο, το πρόγραμμα Infomar. Είναι μια κοινοπραξία μεταξύ ε, του Θαλάσσιο Ινστιτούτου τούτου ε, και καλύπτει 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, των ε, πιο εμπορικών θαλασσίων ουσιαστικά εκτάσεων της ε, Ιρλανδίας. Επίσης ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα βιώσιμο νομικό πλαίσιο μεταξύ των τομέων πολιτικής για να διασφαλίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών. Πολύ συχνά έχω συναντήσει αυτό δυστυχώς ε, και πολύ συχνά και ε, εγώ έχουμε, έχω δει ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ διάφορων πολιτικών. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια και έτσι δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κοινό σκεπτικό μεταξύ των διάφορων φορέων που συμμετέχουν σε αυτού του έτσι ώστε να υπάρχει ένα συνολικό στόχο και όλοι να βλέπουν ποιο είναι ο στόχο και να προσπαθούν να διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου αυτού, παρά ε, να έχουν παροπίδες ε, και να μην διευκολύνουν όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε σαφείς πρακτικούς κανόνους, θαλάσσιο χωροτεξικό σχεδιασμό και σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης παρακτήων ζωνών. Αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν σε διαβούλευση με, τους, ε, με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και αν γίνει αυτό μπορούμε έτσι να αναπτύξουμε περισσότερο το δυναμικό της θάλασσας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε σχέση με διάφορους τομείς. Έχουμε το τομέα της, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πραγματικό ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες με την ολική, υπελογική, κυματική ενέργεια και πρέπει να προωθήσουμε τα κλάστερ ε, προκειμένου να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και πρέπει να υποστηρίξουμε project και πιλωτικά σχέδια που συνεχίζονται μάλιστα σήμερα και επίσης ε, πρέπει να υπάρχουν και συνδέσεις διαδικτύου και ικανότητες ε, διαβίβασης. Πρέπει να συσταθούν όλα αυτά γιατί δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε υπεράκτια, αιωλική, υπεραιωλική, κλιματική ενέργεια κτλ. Ε, φυσικά θα χρειαστούν πολύ μεγάλες επενδύσεις, όμως θα έρθουν οι επενδύσεις αυτές σα είπα, θα έρθουν οι επενδύσει όταν υπάρχει ασφαλεία δικαίου και όταν υπάρχει και βεβαιότητα ότι οι επενδυτές θα διευκολυνθούν στο έργο αυτό. Και φυσικά υπάρχει μαζική ευκαιρία για την Ευρώπη που εξαρτάται πάρα πολύ από την εισαγωγή των καυσίμων από διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι αυτή για μας και πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα για να να αναπτύξουμε αυτό το δυναμικό το συντομότερο. Έτσι, είχαμε και μια σειρά συναντήσεων εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί περάκτια παραγωγή αερίου εδώ στην Ευρώπη θα συνδυαστεί με την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών που εμφανίζονται καθημερινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλο ένα και περισσότερο τα τα αερίου που υπάρχουν στην ανεκτή θάλασσα. Και αν δούμε τις διάφορες ε, μελέτες επιπτώσεων που έχουν γίνει, τις διάφορες αξιολογήσεις, υπάρχει τεράστιο δυναμικό και για την ε, δική μου χώρα, αλλά και για άλλες χώρες υπάρχουν ε, τέτοια κοιτάσματα που δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμη και προτιμώ να έχουμε αέριο που έρχεται από το εσωτερικό της Ευρώπης παρά να το εισάγουμε από μη σταθερά καθεστώτα, από σταθερή καθεστώτα. Είδα το καλλιέργεια είναι άλλος τομέας που είναι ιδιαίτερα ζωτικός. Ε, το 90% των επιχειρήσεων καλλιέργεια είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει που παρέχουν 80.000 θέσει εργασία, αλλά πάνω από τα 2 τρίτα των ε, θαλασσινών ε, που τρώμε στην Ευρώπη, καταναλώνουμε στην Ευρώπη και πάλι εξάγεται από τρίτε, από χώρε. Και πάλι λοιπόν εδώ πρέπει να προσδώσουμε σημασία στην διτοκαλλιέργεια και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίε των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. Έχουμε, παραδείγματο χάρη στη δική μου χώρα, μεγάλε επιχειρήσει ιδιωτοκαλλιέργειας και υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για να δημιουργηθούν μεγάλες ε, επιχειρήσεις δεδοκαλλιέργεια. όμως πρέπει να εξετάζονται αυτές οι αντιρρήσεις γιατί υπάρχουν ε, ανάλογα με τα συμφέροντα των διαφορών ομάδων αποκλίνουσες απόψεις και μερικές φορές μπορεί να σταματήσουν κάποια καλά project έτσι λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να έχουμε επιχειρήματα που να βασίζονται στις ε, επιστημονικές απόψεις γιατί και αυτός ο τομέας ε, έχει τεράστια δυναμική στην Ευρώπη και μπορεί να υλοποιηθεί με έναν τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τώρα, γαλάζια βιοτεχνολογία, ένας άλλος ε, τομέας, ε, σχεδόν ανεξερεύνητος, όμως αποτελεί και αυτός ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Εδώ Επίσης μπορούμε να αναπτύξουμε καλλιντικά, φάρμακα, τεράστιο δυναμικό και εδώ και βλέπω να τονίζετε και να υπογραμμίζεται σε διάφορες συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο και στις τρογγυλές τράπεζες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτήν την τομέα σε πάρα πολλούς ε, σε περιοχές της Ευρώπης και κάτι τελευταίο ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη ε, και στις ε, παράκτες και τις απασχόλησεις στις παράκτες περιοχές δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξη όπως τα θελασσία αθλήματα και επίσης πρέπει να αναπτυχθεί η κατάλληλη υποδομή γιατί δημιουργεί ε, τεράστια δυναμική για την ανάπτυξη του διασυνοριακού τουρισμού θα πρέπει επίση ε, να δούμε και όλε αυτέ τι υπέροχε ιδέε που έχουμε, του αυτοκινητοδρόμου τη θάλασσα και άλλε τέτοιε ιδέε που μπορούν να δημιουργήσουν θέσει εργασία, να αναπτύξουν τη δυναμική τη θάλασσα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο φιλικό προ το περιβάλλον, έτσι ώστε η Ευρώπη να καταστεί πιο ανταγωνιστική από ό,τι είναι και φυσικά για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την ύφεση την οποία βιώνουμε σήμερα και ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πόσο τεράστια είναι η δυναμική στο τομέα αυτό και υποστηρίζουμε το έγγραφο της Κομισιόν και Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ε, και την ασφαλή δικαίου αλλά και τις απαραίτητες υποδομές για τις επενδύσεις για να αναπτυχθεί αυτό το δυναμικό. Επομένως, η γαλάζια ανάπτυξη είναι ο νέος τρόπος ανάπτυξης. Ο κύριος Τριολιέν, παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο ε, που υπογραμμίζει όλα τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτή την πρωτοβουλία για τη γαλαζιανάπτυξη. Η ανακοίνωση αυτή της Κομισιόν απαριθμεί με ακρίβεια μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που μας επιτρέψουν ε, να υποφεληθούμε όσο δυνατόν περισσότερο από τις παράκτη περιοχές. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία και συμπληρώνει το έργο που υλοποιήσαμε γύρω από την ολοκληρωμένη θελάσσια πολιτική. Και να ομολογήσω ότι η Κομισιόν Μάλλον ε, δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι πιο αρμόδια ε, για να μελετήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή γιατί ανέλαβε την κυρία Γνωμοδότη Επιτροπή αυτή δεν το καταλαβαίνω και όχι εμείς. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα να επιμείνω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν ε, κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά πολύ αρνητικά για το περιβάλλον και αυτό παρά το ότι ε, θα έπρεπε να επιβληθεί ένα επιτακτικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, βλέπουμε τις επιπτώσεις από την εδατοκαλλιέργεια, τον τουρισμό, υπάρχουν αρκετά ε, συνέπειες, μία μελιτές και Βεβαίως η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική όπου τίθεται αυτή η πρωτοβουλία για την γαλάζια ανάπτυξη θα πρέπει να απαντήσει σε, αυτό το, σε αυτήν την επιτεκτική ανάγκη συνολικής ε, συνοχής ε, για την προστασία ε, της θάλασσας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος η ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να γίνεται για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες καθώς ε, ο θαλάσσιος χώρος είναι ένας χώρος ε, συνοριακός αλλά και ένας χώρος ανταλλαγής. Η ικανότητα που θα έχει η Ένωση να επιμεριστεί με τους ε, γειτονές της το κόστος αλλά και το όφελος αυτής της, θαλάσσιας, της γαλάζιας ανάπτυξης θα είναι και ένας τρόπος να αξιολογήσει τη θέση της παγκοσμίω στην παγκοσμία σκηνή. Και πάλι λυπάμαι που η παγκόσμια διάσταση της Ένωσης υποτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη, αναφέρθηκαν ε, κάποια στοιχεία εδώ στο κείμενο και μας εξηγούν ε, μέσα φύνεται η δράση των κρατών μελών και της Ένωσης για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι επιχειρησιακά βήματα που υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις περιφέρειες δεν υπογραμμίζονται παρκώς. Και αν η γαλάζια ανάπτυξη καταστεί προτεραιότητα, οι πιλωτικές μας πρωτοβουλίες που επιλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε και αυτές ε, να τονίζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Και όπως υπογραμμίζει αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περιφερειακές ε, περιοχές και άκρως απομακρυσμένες περιοχές έχουν στρατηγικό ρόλο στην γαλαζιά ανάπτυξη. Επομένως, ε, ε, αν προσεγγίσουν οι λέει τον ένας τον άλλον, θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να επωφεληθούν όλοι από αυτή τη στρατηγική. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως αυτές τις προσπάθειες συνοχής της Ένωσης σε ό,τι αφορά τις παράκτη και θαλάσσιες ζώνες. Δυστυχώς ε, ε, δεν ε, μπορούμε να προσυνδέσουμε τη συζήτηση αυτή από το θέμα του προπολογισμού, από τα δημοσιονομικά, γιατί αν δεν υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση, τίποτα από όλα αυτά δεν θα υλοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χρυσόγελος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε τη στρατηγική που βασίζεται στη διαχείριση θαλάσσιων λεκανών, έχοντας υπόψη ότι αντίστοιχα για τους υδατικούς πόρους μιλάμε για τη στρατηγική σε επίπεδο υδρολογικών λεκανών. Όπως ακριβώς για τα θέματα των υδατικών πόρων και η στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες πρέπει να προωθεί τη βιωσιμότητα. Έτσι ώστε πραγματικά να εξυπηρετεί την περιφερειακή ανάπτυξη την ανάπτυξη δηλαδή βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την απασχόληση και ιδιαίτερα την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών χρήσεων του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, να διασφαλίσει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιπικιλότητας, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδομών από φαινόμενα διάβρωσης, πολλές φορές είναι αποτέλεσμα παρεμβάσεων απρογραμμάτιστων ή χωρίς κατάλληλε μελέτε, στην παράκτια ζώνη και βέβαια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων, ρήπανση καθώς και φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Άρα στην, ε, πρέπει να αναπτύξουμε κατάλληλα οικονομικά και διοικητικά εργαλεία που να μπορέσουν να εφαρμόσουν μια τέτοια στρατηγική, βιώσιμη στρατηγική διαχείριση των θαλάσσιων λεκανών. Τώρα, πρέπει πραγματικά να υπάρξει και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών εργαλείων και πολιτικών και είναι σημαντική η πρόταση για ανάπτυξη θαλάσσιων κλάστερς που όμως θα προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών με στόχο όχι μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και τη διασφάλιση της υγείας των θαλάσσιων οικοστημάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και εξασφάλιση θέσεων εργασίας για να είναι αποδεκτά αυτά τα σχέδια πρέπει να είναι και αποτέλεσμα, αποτέλεσμα διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να είναι δηλαδή αποτέλεσμα συστηματικού κοινωνικού διαλόγου και πολύ σημαντικό επίσης να υλοποιούνται μέσα από σχήματα πολυεπίπεδης συμμετοχής διακυβέρνησης. Δηλαδή να μην είναι σχήματα τα οποία κάποιος άλλος έχει αποφασίσει, αλλά να εντάσσεται στη στρατηγική που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή, η πολυεπίπεδη συμμετοχική διακυβέρνηση να είναι πραγματικότητα. Βέβαια, πολλές φορές η στρατηγική αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ε, πολλές φορές οι θαλάσσιες λεκάνες δεν περιορίζονται μέσα στα εθνικά σύνορα, άρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και για τις πολιτικές και για τις στρατηγικές ε, και διασυνοριακά και μεταξύ διαφορετικών περιφερειών. Δηλαδή τα διοικητικά όρια δεν είναι πάντα και οικολογικά όρια, επομένως θα πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Επίσης, για να προωθήσουμε μια τέτοια στρατηγική χρειάζεται και να αναβαθμίσουμε δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να υπάρξουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ε, και στο επίπεδο της τεχνικής και της ε, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνεργασία μεταξύ ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορες χώρες και περιφέρειες, για να μπορέσουν ε, ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, στα νέα προσόντα, στις νέες προδιαγραφές ενός ευραίου φάσματος θαλάσσιων και κυρίως πράσινων θαλάσσιων επαγγελμάτων. Ήδη υπάρχουν ε, αρκετές τέτοιες δραστηριότητες, αλλά χρειάζεται να ενισχυθούν και να δικτυωθούν μεταξύ τους σε επίπεδο ακαδημαϊκό και ερευνητικό. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή έχουμε συζητήσει και στο Ευρωπαϊκό και στο Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν έχει καταθέσει αρκετά εργαλεία, όλα αυτά τα εργαλεία πρέπει να ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται γαλάζια ανάπτυξη, έτσι ώστε πραγματικά να είναι πιο συμβατή με την πράσινη οικονομία. Και αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ε, η οδηγία, οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας για τα πουλιά και τους κοτόπους, ειδικά σε ε, αβαθή νερά και σε παράκτιες ζώνες, ή η εφαρμογή της ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, ή η στρατηγική για την ε, προστασία του κλίματος αλλά και την προσαρμογή ε, σε επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης βέβαια των επιπτώσεων, αυτά πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στρατηγικές ε, διαχείρισης ε, σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών. Και αυτό είναι ακριβώς που θα μπορέσει να δώσει και απάντηση στην ανάγκη νομικής σταθερότητας ενός πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει μακροχρόνια ότι οι επενδύσεις που θα γίνονται θα είναι βιώσιμες από κάθε άποψη, όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική θα υπάρχουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θα είναι γνωστά σε κάθε ενδιαφερόμενο να επενδύσει, είτε αυτό είναι ιδιώτη, είτε είναι μικρομεσαία επιχείρηση, είτε είναι συνεταιρισμό. Μια και η επένδυση σε θαλάσσιε περιοχέ είναι βέβαια κάτι αρκετά πολύπλοκο και σύνθετο. Ε, προφανώς χρειάζεται να υπάρξουν ξεκάθαρα αλλά και βιώσιμα σχέδια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνη, γιατί μιλάμε για επεμβάσει σε πάρα πολύ ευαίσθητες περιοχές και οικοσυστήματα που ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει και σε συγκρούσεις χρήσεων αλλά και σε μεγάλες αλλαγές. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι παρεμβάσει που έχουν γίνει σε πολλέ παράκτιε περιοχέ, από μικρά έω μεγαλύτερα έργα, χωρί κατάλληλη προετοιμασία, που έχουν οδηγήσει σε πολύ σημαντικά προβλήματα διάβρωση παράκτια ζώνη. Στη δικιά μου χώρα, περίπου το 25% ίσως και παραπάνω τη παράκτιας ζώνη βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτία τη διάβρωση λόγω άστοχων παρεμβάσεων στην παράκτια ζώνη, αλλά γνωρίζετε ίσω και την ε, έκθεση που έχει γίνει για τη διάβρωση στην Ευρώπη, που δείχνει ακριβώ ότι η παρέμβαση στο όνομα πιθανά τη δημιουργία θέσεων εργασία ή τη ανάπτυξη έχει προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα που εκ των υστέρων δημιουργούν και μεγάλα κόστη στι τοπικέ κοινωνίε. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό πράγματι για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στη θαλάσσια ζώνη πρέπει να τις αξιοποιήσουμε με βιώσιμο τρόπο ε, να δημιουργηθούν πραγματικά βιώσιμες θέσεις εργασίας αλλά με στόχο να μειώσουμε επίσης και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ρήπων στα θαλάσσια περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε μια στρατηγική σταδιακής απεξάρτησης από τη χρήση ορυκτών καυσίμων γιατί βέβαια δεν μπορεί να θέλουμε ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων και διοξιδίου του άνθρακα και να επενδύουμε όλο και περισσότερο σε εξορίξη υδρογονανθράκων, πετρελαίου, φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή. Τεράστιο δυναμικό για ε, οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας υπάρχει αν συνδυάσουμε τη στρατηγική σε επίπεδο λεκάνης, θαλάσσιας λεκάνης με πολιτικές όπως είναι το πρασίνισμα των λιμανιών και της ναυτιλίας. Ε, η διαχείριση, η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων από κάθε είδους σκάφη αλλά και ιδιαίτερα εάν αξιοποιήσουμε τη στρατηγική Leadership 2020, η οποία προβλέπει και τη δυνατότητα να υπάρξουν συμβάσεις μεταξύ περιφερειών ε, επιχειρήσεων κερδοσκοπικών ή υποπροϋποθέσεις, κερδοσκοπικών αλλά και μη κερδοσκοπικών για την ενίσχυση για την ε, κατασκευή σκαφών τα οποία θα είναι μηδενικής, μηδενικών ρήπων, δηλαδή θα βασίζονται κυρίως σε ανανόσιμες πηγές ενέργειας ή τη βελτίωση της, ενεργητικής, της ενεργειακής αποδοτικότητας των σκαφών. Αυτό είναι, παρόλο ότι μοιάζει ότι μια πολιτική για τη βιομηχανία, είναι πολύ σημαντική και για την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί σε χώρες όπως η Ελλάδα κινδυνεύουμε να μείνουμε από ακτοπλοϊκές συνδέσεις, το κόστος των καυσίμων έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη δυσκολία να είναι βιώσιμες οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ παράκτων περιοχών και νησιών. Άρα μια τέτοια στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, φανταστείτε τα νησιά να μην έχουν συνδέσει ακτοπλοϊκέ. Οτιδήποτε άλλο στάμε δεν είναι εφικτό να προχωρήσει. Υπάρχει λοιπόν τεράστια καινοτομία αν αναπτύξουμε και σκάφη τα οποία είναι πιο πράσινα, αλλά και ένα δίκτυο ε, σταθμών παραγωγής, αποθήκευσης και διανομή ενέργεια που θα βασίζεται σε ανώσιμε πηγές ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε όλη την παράκτια ζώνη. Γνωρίζουμε ότι στη Βαλτική δημιουργείται δίκτυο με σταθμούς από υγροποιημένο αέριο, αλλά αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε κάθε χώρα και επίσης πρέπει να αναλογιστούμε και την κλιματική αλλαγή. Όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν παντού και η παράκτια ζώνη, offshore περιοχές και τα νησιά θα μπορούσαν να, ήταν κάλιστα, να συνδεθούν κάλλιστα στα πλαίσια μιας στρατηγικής θαλάσσιων ε, λεκανών να, να, να αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο παραγωγής, αποθήκευση, διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Και βέβαια ήδη έχουν προχωρήσει ορισμένα προγράμματα σε πιλωτικό κυρίως επίπεδο. Έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα έξυπνα δίκτυα και όχι τα παραδοσιακά δίκτυα για την απασχόληση και νέες μορφές περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, τέλος, δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά, τα θέματα της αλίας και τα θέματα του τουρισμού. Επειδή ε, πριν από λίγο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον Λομέλη αποφασίσαμε για μια νέα στρατηγική για την ε, κοινή, αγροτική, για την κοινή αλληλευτική πολιτική, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό η πράσινη, η, μάλλον η γαλάζια ανάπτυξη, όπως ονομάζεται, να συνδεθεί με βιώσιμες μορφές αλίας. Δεν αγνοούμε ότι υπάρχουν πράγματι σήμερα αναπτυγμένες επενδύσεις ε, στην ηχθιοκαλλιέργεια αλλά αυτό που χρειάζεται να ενισχύσουμε είναι κυρίως βιώσιμες μορφές αλίας, επανάκαμψη της θαλάσσιας βιοπικιλότητας, δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που θα δώσουν τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, κυρίως σε νησιωτικές παράκτιες και απομονωμένες περιοχές, να αποκτήσουν βιώσιμες θέσεις και νέα επαγγέλματα και ταυτόχρονα βέβαια να πετύχουμε στόχους όπως είναι η ανάκτηση της βιοπικιλότητας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κτλ. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση και να το, ταμείο, το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και να δώσει μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του προτεραιότητα και κατεύθυνση σε τέτοιες μορφές δραστηριότητας που θα βοηθήσουν και νέους ανθρώπους να μπουν στο επάγγελμα του ψαρά και νέα επαγγέλματα τα οποία θα βοηθήσουν παράλληλα και στην, και στην επανάκαμψη της βιοπικιλότητας. Τέλος, για τον τουρισμό. Αυτό που χρειάζεται να στηρίξουμε γιατί είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα πολλών περιοχών, είναι οι υπεύθυνε μορφές τουρισμού και η σύνδεση αυτών των μορφών τουρισμού με τους τοπικούς πόρους, την τοπική παραγωγή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνίζεται χαμηλού κόστους προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και πολύ περισσότερο να ενθαρρύνεται η μη διαφοροποιημένη τουριστική ανάπτυξη. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε στα πλαίσια μια τέτοιας στρατηγικής είναι η κάθε περιοχή, η κάθε θαλάσσια λεκάνη, να δει ποια είναι τα πλεονεκτήματά της κοινωνικά, παραγωγικά, ε, περιβαλλοντικά και να βασίσει το μοντέλο της, του τουρισμού ε, σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία, και το μοντέλο αυτού του τουρισμού να διασφαλίζει μακροχρόνια τη διατήρησή τους. Εδώ υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε μορφές τουρισμού που δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα, όπως είναι ο οικοτουρισμός, όπως είναι ο αλλιευτικός τουρισμός, ο καταδυτικός και άλλες μορφές ήπιου τουρισμού του νερού, να μην κάνουμε το λάθος να επεκτείνουμε διάφορες μορφές τουρισμού του νερού που είναι ε, στο τέλος γίνονται και για τις περιοχές, αλλά εκείνες ακριβώς τις μορφές τουρισμού του νερού που διατηρούν μακροχρόνια τα χαρακτηριστικά ε, αυτών των περιοχών που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε ο Φραγκίσκος Αλφόνση. Ναι, σύντομα. Δύο σημεία παραπάνω από αυτά που υπόθηκαν για την έκθεση. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στο συνδυασμό της στρατικής αυτής με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, προτείνουμε ότι θα καταθέσουμε τροπολογία και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε σε ποιο βαθμό θα ήταν καλό και για την πράσινη ανάπτυξη αλλά και για την αντιμετώπιση του θερμοκηπίου, του εφέτου θερμοκηπίου να ληφθούν μέτρα πιο βολονταριστικά, ιδίως για τη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις μας για να προσθεθεί κάτι σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω τις παρατηρήσεις του σκιώδους εισηγητού μας ε, πάνω στο σχέδιο έκθεσης αυτό. Καταρχήν ε, θα ήθελε να επικροτήσει το σχέδιο έκθεσης. Επίσης πιστεύει ότι η θάλασσα και οι ακτές ε, είναι πολύ σημαντικά για, τις, ε, για την οικονομία, αντιπροσωπεύουν το 5% της οικονομίας, ε, το 5% των θέσεων εργασίας και 5 Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνουν και σωστές έρευνες στον τομέα της ενέργειας. Υπάρχει σημαντική ανάγκη να ε, αυξήσουμε το δυναμικό της ε, υπεράκτιας ε, παλιριακής και θαλασσιάς ενέργειας. Έτσι μπορεί να μειωθεί η ανάγκη χρήσης εδαφών στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, Ε, μας ενδιαφέρει ο παράκτιος ε, και ο θαλάσσιος τουρισμός σε, κάποιους, σε κάποιες περιοχές. Ε, ο τουρισμός αποτελεί πηγή πρόσθετου εισοδήματος για τις παράκτιες κοινότητες. Σε κάποιες όμως μειονεκτικές και απόμακρες περιοχές είναι ο μόνος σημαντικός οικονομικός τομέας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει ε, υποδομή στις περιοχές αυτές όπως είναι ε, λιμένες και άλλα, προσελκύοντας ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και η ομάδα μα θα υποβάλει και τροπολογίες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάιτσε Σίμερς ε, είναι παρόν από τη Γενική Διάθεση για τη Θάλασσα. Θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Πολύ σύντομα να πω ότι ευχαριστούμε τον εισηγητή και την Επιτροπή για τις θετικές παρατηρήσεις πάνω στην ε, ε, πρωτοβουλία αυτή. Οι παρατηρήσεις που έγιναν αναφέρονται στη θαλάσσια οικονομία, τη γαλάζια οικονομία. Ε, πολύ σημαντικό είναι το δυναμικό που υπάρχει εδώ και προσπαθούμε όχι να καλύψουμε το σύνολο της θαλάσσιας οικονομίας, αλλά να τονίσουμε κάποιους τομείς όπου μπορεί να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να δημιουργηθεί δυναμικό για την μελλοντική ανάπτυξη ε, και δημιουργία θέσεων απασχόλησης Σημειώσαμε όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική θα προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε αυτά στον προγραμματισμό για τα νέα διαφθορτικά και περιφερειακά ταμεία. Και υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο εδώ που έχει να κάνει με την έρευνα και την χρηματοδότηση της καινοτομίας στο πλαίσιο του Horizon 2020. Επίση, όσον αφορά τη νομική ασφάλεια, πιθανότατα να γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν υιοθέτησε την πρότασή της για οδηγία πάνω στον θαλάσσιο χωροτεξικό σχεδιασμό. Ε, ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει νομική βεβαιότητα για τις εταιρείες ε, που θέλουν να επενδύσουν στη γαλάζια οικονομία. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σον, έχει την τελευταία λέξη άμα θέλει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με ενθάρρυνε πολύ το ότι ήταν συνεπείς οι, οι παρατηρήσεις που έγιναν από τους διάφορους ομιλητές. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εδώ. Ε, θα πρέπει να χειριστούμε το θέμα ξεχωριστά, θα πρέπει να ε, χειριστούμε σωστά την υποδομή και θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες για το περιβάλλον. Όπως είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα αυτά βήμα-βήμα και να επικεντρωθούμε στα θέματα όπου μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα γρήγορα και να προχωρήσουμε στα, στις πιο ακριβές προσπάθειες ε, αργότερα. Οι ομιλητές ε, ανέφεραν ποιες είναι, ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Ε, μάλλον θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσουμε στον τουρισμό αλλά εν ευθέτω χρόνο θα είναι σημαντικές και οι άλλες πρωτοβουλίες. Χάρηκα πολύ που οι βουλευτές τόνισαν τη σημασία ε, εκμετάλλευσης ε, ε, των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να παράγουμε τη δική μας ενέργεια εδώ στην Ευρώπη, αντί να εισάγουμε τόσο μεγάλο ποσοστό από αλλού. Σημειώνουμε ιδιαίτερα αυτό που είπε η Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική ασφάλεια. Και όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία και το ορίζον 2020 στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που τα ακούω αυτά. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Και στο μέλλον νομίζω θα ε, αποδεχθεί ότι πρόκειται η αποφασιστική κίνηση. Ευχαριστώ, Σον. Ε, θα πρέπει να λάβουμε απόφαση σχετικά με την ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Προτείνω 22 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, ως προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα όλους να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να παραμείνουν ε, οι συντονιστές, διότι έχουμε τώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ λοιπόν να αποχωρήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αμέσως τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.